Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ε, καλωσορίσω όλους ε, στην κοινή συνεδρίαση και συζήτηση με την ε, Επίτροπο κυρία Μάλστρομ και τον κύριο Χόγκαν. Από την άλλη σας καλωσορίζω. Θα συζητήσουμε το θέμα των επιπτώσεων Τόσων στη γεωργία που θα έχουν οι συμφωνίες εμπορίου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Αυτή η συζήτηση μας συνοδεύει εδώ και κάμποσο καιρό. Ξέρετε ότι έχουν γίνει κάποιες διαπραγματεύσεις για την TTIP, για την ΣΕΤΑ. Οπότε στο θέμα της γεωργικής πολιτικής βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ε, η σωστή εξέλιξη του εμπορίου και η συνετή εξέλιξη του εμπορίου οδηγεί σε ανάπτυξη, ειδικά ε, στον τομέα της γεωργίας έχουμε αντίστοιχα ανάπτυξη ε, και Βλέπουμε ότι μία έχουμε μία ε, βιομηχανία στην Ευρώπη, βιομηχανία τροφίμων η οποία είναι προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές. Όταν όμως κοιτάμε τον Καναδά μιλάμε για ένα επιθετικό ε, συμφέρον έναντι της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, ειδικά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα τυριά. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα επεξεργασμένα ε, προϊόντα αλλά και για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, βέβαια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίω. Βλέπουμε βέβαια ότι μια πολιτική που είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά προς τις εξαγωγές ε, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα και γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς ε, θα δράσουμε στο μέλλον ε, ανεξάρτητα και από το εμπόριο. Το θέμα λοιπόν είναι ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες οι προκλήσεις. Αυτό θα συζητήσουμε και όπως είπα χαίρομαι που έχουμε εδώ τις δύο επιτρόπους που είναι υπεύθυνε για τα αντίστοιχα θέματα. Έχουμε την εξή ε, σειρά προβλέψει Οι επίτροποι θα αποφασίσουν από μόνο τους ποια θα μιλήσει πρώτη. Οπότε βλέπω ότι ε, έχουμε εδώ τον συνάδελφο ο οποίος θα θέλει πρώτος να μιλήσει πριν τις επιτρόπους. Okej. Ο κύριο Σεκέρσκι, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους επιτρόπους και τους συναδέλφους στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Ε, είναι ιστορική σημασία σε αυτή η κοινή συνεδρίαση, εξαιρετικά σημαντική και για την κατάσταση και λόγω της κατάστασης ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν εξαρτάται μόνο από την κοινή γεωργική πολιτική, δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος του γεωργικού προϋπολογισμού, αλλά η Ευρωπαϊκή Γεωργία εξαρτάται και από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Και μάλιστα το λέω αυτό με κάποια πικρία, γιατί θεωρώ ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και στις ε, επιτροπές ε, που ασχολούνται με εξωτερικά θέματα, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, δυστυχώς ανεπαρκώς λαμβάνονται υπόψη, και το λέω αυτό με πικρία, ανεπαρκώς λαμβάνονται υπόψη οι οι συστάσεις και απόψεις της Γεωρικής Επιτροπής για το πώς επηρεάζουν οι εξωτερικές διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Εγώ πολύ συχνά ε, μίλησα και μιλάω για αυτή τη σημασία των εξωτερικών παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και δεν θα κουραστώ να το λέω γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξωτερικές διαστάσεις εξού και η σημασία που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες και εμπορικές διαπραγματεύσεις γιατί επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Για πολλά θέματα και για τις γεωργικές τιμές, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Πολύ συχνά, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, δυστυχώς παραμελούνται τα γεωργικά θέματα προς όφελος άλλων κλάδων, της βιομηχανίας, των χρηματοπιστωτικών θεμάτων και θύμα στο βωμό των άλλων κλάδων είναι η γεωργία. Ενώ εμείς έχουμε επαφές με τους γεωργούς και με εκπροσώπους του αγροεπιστηστικού τομέα, που είναι ένας ευρύτατος τομέας. Ε, δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργία ε, ή μόνο στη μεταποίηση ή μόνο στο εμπόριο. Είναι ένας ευρύτατος τομέας της παραγωγής. Αυτός που καλύπτει τη γεωργία και τα μέσα της γεωργίας. Και επίσης έχουμε πολλούς παράγοντες στην αγορά, πολλές επιχειρήσεις ε, που και αυτές επηρεάζουν την γεωργική ανάπτυξη μέσω των εμπορικών τους συμφωνιών και πρακτικών. Ε, πολλές αποφάσεις λαμβάνονται όχι σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η εμπορική διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική και επηρεάζει και τις περιφερειακές συμφωνίες. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε ιδιαίτερος για να αναδείξουμε τη σημασία που έχουν όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες στη γεωργία και να καταδείξουμε το σωρευτικό αποτέλεσμα που έχουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις και εμπορικές συμφωνίες στη γεωργία. Η ΣΕΤΑ, η συμφωνία Μερκοσούρ, η διαπραγματεύσει του TTIP, οι εμπορικέ διαπραγματεύσει με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όλε αυτέ οι εμπορικέ διαπραγματεύσει ε, εμπεριέχουν δυνάμει απειλέ για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και αυτέ οι απειλέ είναι πολύ σημαντικέ κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόταση για την κοινή αυτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Διεθνού Συμπορίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και τους επιτρόπους που είχαν την καλοσύνη να έρθουν για την συζήτηση αυτή γιατί περιμένουμε πραγματικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις τους για αυτό το σημαντικό τομέα των ε, επιπτώσεων στη γεωργία που έχουν οι εξωτερικοί παράγοντες, η εξωτερική διάσταση. Γιατί γνωρίζουμε πώς επηρεάζουν οι εξωτερικοί παράγοντες τις τιμές των γεωργικών προϊόντων, αλλά και πόσο σημαντική είναι η γεωργία για τον κόσμο. Και ε, πολλές τρίτες χώρες προσφέρουν ιδιαίτερη προστασία στην τοπική τους γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Συμπροάντρε. Έχει αποφασίσει μια μήπως η Επιτροπή. Ωραία. Αποφασίσαμε να ξεκινήσει η κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο με την Ίντα, την οποία συναντώ συχνά, αλλά και την Επιτροπή Άγκρη και αυτό εκφράζει την συνεργασία που έχουν οι ομάδες μας ε, στη Συμφωνία Συμπηρία και είναι λοιπόν πολύ καλό το ότι συναντώμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζω ότι όλοι ενδιαφέρεστε για τις ε, εμπορικές συμφωνίες ε, και όλοι έχετε ασχοληθεί με αυτό. το TTIP, το σέτα, καθώς βρίσκεται και όλες τις άλλες συμφωνίες με την Ισία και ούτω καθεξής και είναι χαρακτηριστικό ε, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ευημερίας, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά φροντίζουν την επιστημιστική μας ασφάλεια, ασφάλεια αλλά και την αγροτική μας ταυτότητα και γι' αυτό το λόγο η γεωργία πάντοτε εφορούσε κάτι παραπάνω από τα οικονομικά αλλά όλες τις υπόλοιπες αξίες μας και αυτό αντικατροπίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τις εμπορικές συμφωνίες. Στόχ, πρώτος στόχος είναι οι ανοιχτές αγορές, τους ώστε να δημιουργηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για τους επενδυτές, τους επιχειρηματίες, τους καταναλωτές, του Ευρωπαίου, αλλά θεωρούμε ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι και κομμάτι των ε, αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμπεριλαμβάνονται και σε άλλες πολιτικές όπως είναι η επιστημιστική ασφάλεια. Και αυτό είναι η βάση των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την Γεωργία και όλα υποστηρίζουν ε, την ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνίες όσον αφορά τις, τα, τα γεωργικά προϊόντα αλλά και την πρόσβαση σε νέες αγορές. Εμείς βέβαια έχουμε προσαρμοστεί σταδιακά με το χρόνο και σήμερα η ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις ε, επιθετικές αλλά και αμυντικές ανησυχίες έχει ε, αλλάξει. καταργούμε δασμούς, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για τα προϊόντα μας. Πέρσι ο τομέας είχε ένα θετικό εισιζύγιο και 8% έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια το ε, εμπόριό μας, το οποίο σημαίνει ότι δείχνει ότι αυτό είναι καλό γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ανέρχονται στα 1,4, ε, υποστηρίζουν 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ήπειρο και πέρσι οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αντιστοιχούσαν στο 7% όλων των εξαγωγών και ο ρυθμός αυτός αυξάνεται ετησίως. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του αγροτικού ε, τομέα όπω και του υπόλοιπου τομεί θα πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να προσεγγίσουμε νέε αγορέ και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται νέε εμπορικέ συμφωνίε. Χρησιμοποιούμε αυτέ τι συμφωνίε για να ξεπεράσουμε τρία εμπόδια. Πρώτον φυσικά την, τα εμπόδια, ε, τα κλασικά εμπόδια όπως είναι οι δασμοί. Πολλοί λένε ότι δεν έχουν απομείνει πολλοί δασμοί και υπάρχουν αρκετά εμπόδια για τις αγροτικές εξαγωγές και η τελευταία έρευνα για την ε, σορευτική επίπτωση των εξαγωγών έδειξε ότι στις 12 ε, εταίρους ε, ε, ελεύθερου εμπορίου ανέρχεται στο 45% για τη ζάχαρη στο 20%, 35% για το κρέας. Στην περίπτωση του Καναδά τώρα οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν δασμούς της τάξης 10 με 25% όμως μέσω του ΣΕΤΑ μπορούμε ε, να μειώσουμε κατά 29% τους δασμούς, το οποίο σημαίνει όλα τα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Αλλά και στα πιο ευαίσθητα προϊόντα ε, του Καναδά έχουμε τη δυνατότητα να διπλασιάσουμε τις εξαγωγές μας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συμφωνία που έχουμε με το Βιετνάμ. Εκεί η αφαίρεση των δασμών ε, τα ε, κρασιά, τα υνοπνευματόδη, ε, τα ε, προετοιμασμένα γεύματα, αλλά και στην Ιαπωνία εκεί η αντιστοιχεία είναι κάτω από το 35% και μπορούμε να φτάσουμε το 500%. Οπότε μπορούμε να έχουμε μια σημαντική βελτίωση για προϊόντα όπως είναι το χοιρινό, τα γαλακτοκομικά Καθώ επίσης και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι τα ζαχαρωτά, η σοκολάτα, τα ζυμαρικά και γι' αυτό συζητάμε με τους συναδέλφου στην Ιαπωνία. Ακόμα και με εταίρου στη Μερκοσούρ θα πρέπει να επικεντρωθούμε Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ε, για τα γαλακτομικά, χοιρινά, ε, το λάδι, υπάρχει δυνατότητα για μεγάλο κέρδος σε περίπτωση που καταργηθούν οι δασμοί. Όμως αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης ε, τα εμπόδια τα οποία αφορούν τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα για να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε λαμβάνουμε υπόψη το δικαίωμα της ε, κάθε κυβέρνησης να νομοθετεί, υπερασπιζόμαστε αυτό το δικαίωμα στην Ευρώπη, αλλά και στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας. Οι κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουν την ευαισθητική ασφάλεια και να προστατεύουν το περιβάλλον. Όμως ε, δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο ότι ε, υπάρχουν αγνές προθέσεις παντού. Πολύ συχνά οι κανονισμοί αυτοί καταπατώνται, οπότε είναι δυνατό να έχουμε πιο αποτελεσματικά ε, αποτελεσματικές μεθόδους μέσω ε, των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε τους νομοθέτες και από τις δύο πλευρές και να διευκολύνουμε τη διαδικασία εξέβρεσης λύσεων. Για παράδειγμα, το ζήτημα του ε, αγελαδινού κρέατος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα διαπραγματεύσει μας επέτρεψαν βελτίωση σε συστημικά ζητήματα όπως, η, ε, όπως το, η περίπτωση της περιφερειακής προσέγγισης για ε, για παράδειγμα. Και στο ΣΕΤΑ επίσης ε, οι συμφωνίες που έχουμε με τον Καναδά, οι κτηνοτροφικές συμφωνίες, συμπεριλαμβάνονται στην όλη διαδικασία με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαδικασία για ε, έλεγχο φυτών και ε, ζώων και τροφίμων. Ε, η επόμενη, το επόμενο ζήτημα είναι η διασφάλιση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων. Ε, το ε, σκοτσέζικο ουίσκι, το ροκφόρ και ούτω καθεξής και γι' αυτό το λόγο ε, η συμφωνία με τον Καναδά καλύπτει 145 με την Κορέα 160 και 169 με το Βιετνάμ και οι συμφωνίες με τη Σιγκαπούρ, την Κεντρική Αμερική την Νότια Αφρική και εκεί έχουμε μεγάλη βελτίωση και αυτό είναι σημαντικό διότι οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων ανέρχονται το 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τεράστιο ποσό. Βέβαια για να τα πετύχουμε όλα αυτά θα πρέπει να δώσουμε και εμείς κάτι σε αντάλλαγμα. Και αυτό είναι όλο ο σκοπό των διαπραγματεύσεων. Για κάποιε χώρε το βασικότερο κίνητρο μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την πρόσβαση στην ενιαία αγορά για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίε. Όμω κάποιε θέλουν και πρόσβαση στα αγροτικά προϊόντα. Και εδώ είναι ευαίσθητη η κατάσταση διότι αυτά είναι τα πιο προστατευμένα. Και αυτό είναι κατανοητό από τη δική του άποψη διότι πολλοί εταίροι έχουν λίγα ε, αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά για τους ίδιους. Οπότε πώς μπορούμε να το εξισορροπήσουμε αυτό. Υπάρχουν δεσμεύσεις για την προστασία των ίδιων προϊόντων. Το κάνουμε αυτό με περιορισμένη ε, πρόσβαση ε, με δασμολογικές ποσοστώσεις και αυτές οι ποσοστώσεις βασίζονται σε αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στους τομείς που μας απασχολούν και γι' αυτό το λόγο ε, δεν διακινδυνεύουν ε, τα προστοζήν διαφορών αγροτών. Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές προϊόντων που είναι ευαίσθητα για εμάς και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Μερκοσούρ με το αγελαδινό κρέας αυτή η εταίρη λοιπόν είναι πολύ σημαντική για εμάς και όσον αφορά τη γεωργία, όμως δεν πρόκειται να κάνουμε δεσμεύσεις που ξεπερνούν ε, τα όσα αντέχει αυτός ο ευαίσθητος τομέας. Η έρευνα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα και στην οποία θα μπει σε λεπτομέρειες ο κύριος Χόγκαν εξετάζει ε, την επιρροή των συμφωνιών ελευθέρου, ελεύθερου εμπορίου που δημοσιεύθηκε φέτος και δείχνει ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί. Αν εξετάσουμε για παράδειγμα την Κορέα μπορούμε να δούμε ότι ε, το 2011 και έκτοτε οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 40% και ιδιαίτερα στα πιο επεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι τα ζυμαρικά και άλλα, αλλά και ε, τα ε, γαλακτοκομικά κατά 30% και το, και το κρέας κατά 50%. Τα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα δείχνουν ότι ο τομέας θα επωφεληθεί από το σενάριο που εξετάσαμε και αναμένουμε βελτίωση ε, στους τομείς κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων όπου φαίνεται μια πρώτη βελτίωση. Δείχνει επίσης ότι ίσως να υπάρχει ανησυχία για άλλους τομείς όπως είναι το ε, χοιρινό κρέας, το οποίο μας ανησυχεί και θα πρέπει να βελτιώσουμε το έργο μας καθώς προχωρούμε. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι τα οικονομικά μοντέλα μπορούν να δώσουν μια, μονάχα μια περιορισμένη εικόνα. Η έρευνα ε, δεν αποτελεί πρόβλεψη του τι θα συμβεί, διότι οι προβλέψεις ε, είναι δύσκολες, ιδιαίτερα για το μέλλον και καθώς συγχαίρουμε τους συγγραφείς της συγκεκριμένη έρευνα για την πολύ καλή δουλειά τους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί διότι δεν δείχνει ε, το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε ε, τους ε, δασμούς καθότι δεν υπάρχει ένα μέτρο μέτρησης αλλά και όσον αφορά τα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα και εκεί υπάρχουν δυνατότητες δεν έχουμε αναλύσει όμως ε, ζητήματα όπως είναι τα κρασιά, το κρέας που απαρτίζουν το 70% των εξαγωγών μας, ούτε και έχουμε ένα μοντέλο για το πώ επεξεργαζόμαστε τα ευαίσθητα ε, προϊόντα, ε, όπου απαιτείται μεγαλύτερη απελευθέρωση. Και φυσικά είναι μια σημαντική έρευνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήδη έχουμε αρχίσει να την εξετάζουμε λεπτομερώς, όμως έχει παρόλα αυτά κάποιους περιορισμούς. Παρόλα αυτά χαίρομαι να το συζητήσω όλο αυτό, καθώς επίσης και άλλα ζητήματα γεωργικού ενδιαφέροντος αζήτηση σας και σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάνστρομ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Χόγκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Μάστρο, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την εισαγωγή. Αυτή η συζήτηση πιστεύω ότι είναι και αναγκαία και επικαιρή. Ο μελλοντικό ρόλος του εμπορίου στην πολιτική μας ζωή και στην οικονομία είναι θέμα συζητήσεων. Τα εκλογικά αποτελέσματα στον Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ απίτησαν μία συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις του εμπόριου. Και αυτές οι συμφωνίες του ελεύθερου εμπόριο ευκολύνουν την κοινωνία μας και είναι καλή στιγμή που ε, δημοσιεύεται η έκθεση αντικτύπου. Και μπορούμε να δούμε και πόσο γενικό τομέα θα επηρεαστεί από μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε. Τώρα, σαν αφετηρία, επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτά που η Επίτροπο η κυρία Μάλτρο μου είπε, υπενθυμίζοντα ότι το εμπόριο ήδη εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή γεωργία και το τομέα των τροφίμων και υπηρετεί τι τομεί αυτού καλά ε, Ισχυρέ επωφελεί συμφωνίε με του εμπορικού μα εταίρου είναι ο κινητήρα για την ανάπτυξη του τομέα των τροφίμων και των ποτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να είναι υπέρ μα το εμπόριο. Οι διεθνεί αγορέ γίνονται όλο και περισσότερο βασικέ, σημαντικέ για τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισοδημάτων των γεωργών. Όπω είπε ο Επίτροπο Μάλστρομ, η Ανακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπόριο για Όλου τόνισε πόσο φιλόδοξου στόχου έχουμε θέσει. Οι εξαγωγέ αυξήθηκαν κατά 5,7% το 2015 στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο δυναμική που έχει άμεσα αντίκτυπο στον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και στην Ήπεθρο. Το πρώτο ενάμινο ενεστώτο έτου επιβεβαίωσαν αυτή τη θετική τάση και χρειαζόμαστε ένα νέο ρεκόρ στον τομέα εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Φέτο το Σεπτέμβριο σπάσαμε το ρεκόρ. Οι εξαγωγέ έφτασαν μηνιαίο, μηνιαία τιμή περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ. Ξεπέρασε το Σεπτέμβριο του, των παρελθόντων ετών περίπου κατά μισό δι ευρώ. Οπότε η εξαγωγική ε, αξία πήγε 2,2 δις για το χείριο, το 21% αύξηση συγκριτικά με ένα χρόνο πριν και τα νοπά λαχανικά 480 εκατομμύρια ευρώ που είναι μια αύξηση 18%. Αυτό έχει σημασία διότι γνωρίζουμε ότι για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ ε, εξαγωγές έχουμε 14.000 εργασίες που δημιουργούνται. Πρόθεση εξαγωγών προ την Κίνα, πιο συγκεκριμένα, ήταν στο επίκεντρο τη ανακάψεω τη αγορά του χείριου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αντική συνέπεια του εμπάργκο τη Ρωσία για το προϊόν αυτό του χείριου κρέατο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο αγωγέα γεωργικών και προϊόντων και ε, από τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε μάλιστα και έτσι συμβάλλει στην ε, παγκόσμια ανάπτυξη. Πρακτικά αποτελέσματα στην έκθεση δείχνουν ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε πώ μπορούμε να βασιστούμε σε επιτυχίε και να προχωρήσουμε παραπέρα. Είναι μια μελέτη που εδράζεται επί προσωμιώσεων που έγιναν ε, μέσω δύο μοντέλων. Το ένα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών στη Σεβίλη, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Ίδιο αργόριθμο που χρησιμοποιεί ο ΣΑΕ και η ΦΑΟ για την ε, τήσια εικόνα για την παγκόσμια κατάσταση για τη γεωργία στον κόσμο. Δύο θεωρητικοί τα εμπορικά σενάρια εξετάσαμε. Το πρώτο είναι το πιο φιλόδοξο ενδεχόμενο, δηλαδή η απελευθέρωση του εμπορίου για 98,5% των προϊόντων και μερικέ περικοπέ δασμών 50% στα υπόλοιπα προϊόντα που θεωρούμε ότι είναι ευαίσθητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, πιο συντηρητικό σενάριο που εξετάζουμε είναι πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου για 97% των προϊόντων και μερική περικοπή κατά 25% των δασμών για τα υπόλοιπα ευαίσθητα προϊόντα που είναι το 3%. Οπότε η μελέτη συμπεριλαμβάνει μια σύγκριση τη καταστάσεω, δηλαδή ποιο τι θα συνέβαινε εάν ίσχυαν αυτά τα δεχόμενα το 2025 υποθέτοντας ότι και οι 12 συμφωνίες συμπεριλαμβάνονται με την προοπτική που κάνει για το 2025 η Γενική Διεύθυνση Εργία. Για λόγου αφήνεια λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι 12 συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου ε, που αναφέρονται στην ε, Ένωση είναι μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω, Αυστραλία, Καναδά, Ινδονησία, ε, Ιαπωνία, Μερκοσούρ, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππινών, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Ηνωμένων Πολιτειών. Η μελέτη είναι πολύ καλή δουλειά που έγινε. Ένα εξάμεινο χρειάστηκε. Έγινε προβληματισμό όσον αφορά την ανάλυση. Είναι αξιόπιστη ανάλυση, αλλά δεν είναι πρόβλεψη. Ούτε Είναι πρόβλεψη των πιθανών αποτελεσμάτων τη σύναψη των 12 ε, συμφωνιών. Τα εμπορικά σενάρια που διερευνούν ε, τι γίνεται με την απελευθέρωση των δασμών δεν εξετάζουν τι γίνεται με τα συνέπεια μη δασμολογικών μέτρων και, ποια, και ποιες είναι οι παραχωρήσεις να φάσεις ποσοστώσεις, κυρίως για τα προϊόντα, όπου εκεί έχουμε αμυντικά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ήταν αδύνατο να προβλεφθεί για όλε τι εμπορικέ διαπραγματεύσει για προϊόντα και ενδεχομένως θα είχαμε τον κίνδυνο να αποκαλύψουμε στου ομολόγους μας μυστικά μας όσον αφορά τη διαπραγματευτική μα θέση. Η μελέτη καλύπτει λοιπόν όλα τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα και σε κάποιε περιπτώσει όμω σε μαδοποιημένο επίπεδο. Τα μοντέλα δεν επιτρέπουν λεπτομερή αποτελέσματα σε κάποια σημαντικά προϊόντα όπω ανέφερε η Επίτροπο κ. Μάλστρομ. Αλλά παρουσιάζονται λεπτομερή αποτελέσματα για κάποια σημαντικά γεωργικά πρωταρχικά προϊόντα όπω είναι το μπόιο κρέα, χείριο κρέα, γαλακτοκομικά προϊόντα, ζάχαρη και λοιπά. Για τα κατακτικά προϊόντα και το χείριο τονίζει η έκθεση πάρα πολύ καλέ προοπτικέ με σημαντικό ενδεχόμενο ανάπτυξη εξαγωγέ ε, για την παραγωγή και τιμέ παραγωγών για το τυρί που είναι βασικά προϊόντα. Οι συνολικέ εξαγωγέ θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά ένα τρίτο. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο μια αύξηση 9% στις τιμές. Όσον αφορά αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, οι εξαγωγέ θα μπορούσαν να βελτιώσουν τιμέ κατά 16%. Επίση, θετικέ ενδείξει έχουμε για το χείριο κρέα με την ανάλυση που δείχνει τη σημασία που έχει να έχουμε μεγαλύτερη πρωτοσημιακή θέση στην Ασία. Πιο ισχυρή θέση. Είναι υποφελέ και για η συμφωνία κυρίω για το ΣΥΤΟ, η Δημητριακά και για τα πνευματόδη ποτά και τον Ίνο. Η μελέτη δείχνει ότι είναι ευάλωτο ο τομέα του βοηού κρέατο. Δείχνει το μοντέλο μια μείωση στι τιμέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη παραγωγή μακροπρόθεσμα στο βόλιο κρέα. Ε, βλέπουμε και κερδίζει ευαίσθητο τομέα, κυρίω όσον αφορά τι διαπραγματεύσει με του ασιάτε εταίρου μα, που λερικά πρόβιο κρέα και ζάχαρη ίσω να έχουμε μεγαλύτερε εισαγωγέ και επηρεάζεται και το επίπεδο παραγωγή και μέσα έτσι. Για όλα τα ευαίσθητα προϊόντα μα λοιπόν, οι εισαγωγέ ε, για πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, να βάλουν ποσοστό στι αγωγέ είναι σημαντικό και για τα ποροκυπευτικά και λαχανικά είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα. Είναι σαφέ ότι η μελέτη μα δίνει ένα επιχείρημα για μια καλή συμφωνία για το μέλλον, μια κοινή εγωτική πολιτική ισχυρή για το μέλλον, πολύ σημαντική για να διατηρήσουμε τι ειδικέ επιδόσει των διαφόρων τομέων μα, κυρίω τη γεωργία και των τροφίμων και όπω είπε η κυρία Μάλτρομ, να εξασφαλίσουμε βιώσιμη παραγωγή, περιβαλλοντική προστασία και πρακτικέ που αντέχουν στι αλλαγέ του κλίματο. Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διάφορα προβλήματα συνδέονται με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να ενθαρρύνει την καινοτομία για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και περισσότερη καλύτερη αξία για τον γεωργικό τομέα. Ο τομέα ο γεωργοτροφημικό θα ωφεληθεί σημαντικά στην Ευρώπη από την τιμή που αυξάνεται από την άμεση ε, προστασία οι διμερεί συμφωνίε μα δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουμε διάφορα προβλήματα ε, ε, φραγμών ε, που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και να έρθουν. Και συμφωνώ λοιπόν με την Επίτροπο την κυρία Μάλστρομ που ισχυρίζεται ότι τα θέματα αυτά των φραγμών των δεσμολογικών χρησιμοποιούνται για πολιτικού σκοπού και όχι για προστασία των τροφίμων και έτσι παρεμποδίζεται το εμπόριο. Ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπιστούν τα θέματα να αντιμετωπίσουμε απευθεία και αμέσω να συνομιλούμε με του αμέσου εταίρου μα όπω το κάνουμε σε αυτέ τι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου και αυτό το έκανα σε πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια των διαφόρων αποστολών που έκανα σε διάφορες χώρες στον κόσμο το 2016. Και είδαμε κάποιες επιτυχίες ε, όσον αφορά του φραγμούς ε, για το εμπόριο με τους εμπορικούς μας εταίρους. Θα ήθελα ακροθυγώ σε πρώτε προσπάθειε να έρθουν οι μη δεσμολογικοί φραγμοί για το εμπόριο. Μετά το εμπάργκο τη Ρωσία, η Επίτροπη Μάστρομ και Ανδρουκάητη και εγώ αυξήσαμε τι προσπάθειε που καταβάλαμε για να πετύχουμε συγκεκριμένα και ταχεία αποτελέσματα και πρόοδο όσον αφορά μη δεσμολογικού φραγμού και κυρίω όσον αφορά τα θέματα SPS επιδιώξαμε, συνεχούμε για την υγεία και τα φυτογενεμικά και προχωρήσαμε όσον αφορά τι διμερεί διαπραγματεύσει και αυτό στα πλαίσια των αγροτροφημικών μα αποστολών. Επισκέφθηκα το Μεξικό, την Κολομβία, την Ιαπωνία, την Κίνα, το Βιετνάμ και την Ινδονησία και κάθε φορά έφερα μια αντιπροσωπεία του αγροτροφημικού τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και έδωσαν καρπού αυτέ οι προσπάθειε. Εκείνα, παραδείγματο χάρη, ε, ε, τι φραγμού όσον αφορά το βόλιο κρέα και το χείριο κρέα και γενετικό υλικό από τέσσερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά παρόμοια πρόσβαση και από τα άλλα κράτη-μέλη. Η Ιαπωνία έχει άσει την απαγόρευση εισαγωγή βοήου από 7 κράτη-μέλη και η Ολλανδία μπορεί να εξάγει ε, μοσχαρίσιο κρέα ε, και θα ανοίξει ε, η Ιαπωνία καλύτερα να ανοίξει και άλλε χώρε μέλη. Στην Κολομβία είχαμε μακρά διοικητική διαδικασία για τα προκυπηστικά εκεί και κρατάει ένα με δύο χρόνια η διαδικασία και τώρα έχουμε πάει στους δύο μήνες ε, την τελευταία περίοδο και έτσι ε, διευκολύνονται οι από το Βέλγιο. Η επόμενη επίσκεψη αυτού του είδους προγραμματίζεται για τον Καναδά τον Μάιο του 2017 ε, θεωρώ ότι αυτέ οι επισκέψει αποτελούν μια ευκαιρία για συζητήσεις στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, ούτω ώστε να ανοίξουμε τι αγορέ και να δημιουργήσουμε ευκαιρίε για όλε τι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδη, παραμένω πεπισμένο ότι το εμπόριο είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του αεροτροφημικού τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπω είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ συμβάλλει ε, στο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάπτυξη και θέσει και πέρα από τι διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε, εμεί δραστηρία θέλουμε να, έχουμε, να πετύχουμε ισότιμε συνθήκε εξαγωγή και, ε, και μέσω μέτρων πρόθεση να βελτιώσουμε τι εξαγωγέ του αγροτροφωμικού τομέα και για τα φυτογενομικά να μειωθούν οι διάφοροι φραγμοί. Θέλουμε να διευρύνουμε τι δυνατότητε, να ανοίξουν οι βασικέ ε, αγορέ και να επεκτείνουμε το εμπόριο. Επίση, να υπενθυμίσω ότι δηλωμένο στόχο τη υφιστάμενη συμφωνία είναι να προωθήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη, υπεύθυνη διαχείριση των ε, πρώτων υλών και καλή διακυβέρνηση σε διεθνέ επίπεδο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι συμφέρον να διατηρήσουμε το διεθνέ μα εμπορικό θεματολόγιο, να μην χάσουμε το μερίδιο τη αγορά που έχουμε τώρα έναντι των ε, αντιπαλών αλλά να συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέε δυνατότητε για να παράγουμε δυναμική εξαγωγική ανάπτυξη ανάπτυξη μέσω εξαγωγών στον αγροτροφημικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, κύριε Χόγκαν. Περνάμε τώρα στη συζήτηση γιατί είχαμε πολλές ε, πληροφορίες και σαφή κατεύθυνση για τη συζήτηση. Οι συμπρόεδροι συμφώνησαν με την εξή διαδικασία. Θα έχουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και από τις δύο επιτροπές θα ακούσουμε τις απαντήσεις των επιτρόπων και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος για τους λοιπούς ε, ευρωβουλευτές με το σύστημα ε, ερωταπαντήσεων, ping-pong, ε, μία ερώτηση από την Επιτροπή, τα μία ερώτηση από την Επιτροπή Γεωργίας και το βασικό είναι η τήρηση του χρόνου αγόρευσης που είναι 1,5 λεπτό για όλους και θα είμαστε πολύ αυστηροί στην εκτέλεση αυτού του κανόνα. Με το που θα ολοκληρωθεί ο γύρος με τους συντονιστές θα δούμε πόση ώρα θα έχει μείνει. Πάντως, αν θέλετε να ακούσουμε όσο το δυνατό περισσότερο συναδέλφους γίνεται και να γίνει πλούσια συζήτηση, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ αυστηροί στην τήρηση του χρόνου. Για τον πρώτο γύρο λοιπόν, έχουμε 16 συντονιστές, 16 τον αριθμό. 8 από κάθε επιτροπή. Μπορεί να μην θέλουν όλοι να μιλήσουν, αλλά μπορεί και να θέλουν. 1,5 λεπτό στο καθένα λοιπόν. Ο κύριος Βαγουένσα από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Εξεπλάγει που μου δώσετε πρώτα το λόγο. Με ευνηδιάσατε. Σας ευχαριστώ πάντως. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για αυτή τη μελέτη που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι στο μέλλον ε, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Και η μελέτη δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες που εφαρμόζονται προσωρινά. Ακόμη και αν μιλά για ε, απελευθέρωση του εμπορίου για τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, η εις βάθος περιεκτική συμφωνία με την Ουκρανία. Η συμφωνία αυτή με την Ουκρανία προβλέπει ότι η ετήσια αύξηση TRQ για την πενταετία είναι δεδομένη. Γιατί λοιπόν δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη σας και αυτή η συμφωνία με την Ουκρανία για να καθορίσετε αυτά τα σημεία αναφοράς και την πρόσβαση στα γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένων κλάδων, ιδιαίτερα για τις γειτονικές χώρες όπως είναι η Πολωνία που είναι η γειτονική της Ουκρανίας. Αναφερθήκατε και οι δύο ε, την επίπτωση που έχουν οι φραγμοί των υγειονομικών και φυτογειονομικών μέτρων, SPS, στη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων ε, των υγειονομικών φυτογειονομικών ε, μέτρων, γιατί επηρεάζουν τα φυτογειονομικά και υγειονομικά μέτρα πολύ περισσότερο και πολύ πιο αρνητικά τις εξαγωγές από ό,τι οι δασμοί. Τώρα ο Αλμπερτές, ο συντονιστής του ΕΛΚ από την Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ τους ε, δύο συμπροέδρους ε, για το γεγονός ότι έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Η ΕΛΚ, το ΕΛΚ καλωσορίζει και τους δύο επιτρόπους. Ε, ελπίζω να αισθάνεστε καλά μεταξύ μας. Είμαστε μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ και έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θέλουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσα η γεωργία Φύγετε ε, από αυτό το θέμα. Ε, κατά πόσο είναι προς όφελός της. Ε, έχουμε τα καλύτερα προϊόντα. Από το 2003 έχουμε ξεκινήσει με τα καλύτερα τριγιά, τα καλύτερα κρέατα, να, καλύτερα κρασιά, να ανοίγουμε τις αγορές της Αμερικής. Δεν έχουμε λοιπόν φόβο γι' αυτό, αλλά για τους όρους ε, ε, φοβάμαι για το γεγονός ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο μαρτύριο για τους ε, Ευρωπαίους διότι δεν έχουμε πλέον δασμούς. Έχουμε ας πούμε προϊόντα από χώρε που δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μέσα και ο ανταγωνισμός δεν είναι θεμητός. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 είχαμε συζητήσει το θέμα του Μερκόσουρ και είχαμε λάβει σημαντικά ε, μέτρα. Είπαμε ότι με 500 ψήφες υπέρ ότι μόνο όταν τηρούνται συγκεκριμένα στάνταρ για την προστασία των ζώων και των ε, ε χρήσωστών μέτρων θα επιτρέψουμε αυτή τη την ε, συνεργασία. Επόμενος ο συντονιστής ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Προέδρη, ευχαριστώ και τους Επιτρόπους για αυτή τη σημαντική συζήτηση που δεξάγεται σήμερα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε για εκμήγομη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εξαγωγέας σε παγκόσμιο επίπεδο των αγροτροφημικών προϊόντων και απέχουμε πόρο από τη ΣΥΠΑ ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και σε απόψει παρουσίασαν οι επίτροποι. Χρειαζόμαστε λοιπόν το διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη με την οποία αποκτά θέσεις ε, κατακτά την αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι πρωταγωνιστούμε και δημιουργείται, δημιουργούνται ευκαιρίε για τους, τις εταιρείε του τομέα. Όμως πρέπει να πληρούνται προποθέσει όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι ένα ε, από τα κεφάλαια στι διαπραγματεύσει που προωθείται από του διαπραγματευτέ. Σε, σε κάποιου τομεί έχουμε τη συμφωνία με τον Καναδά, σημαντικά αποτελέσματα. Πάνω από 170 γεωγραφικέ ενδείξει αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των εξαγωγών τη Ευρώπη προ τη χώρα. Ε, είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα για τον Καναδά να μπορεί να επιτευχθεί και σε άλλε σημαντικέ διαπραγματεύσει που διεξάγονται τώρα. Ευχαριστώ. And for... από την Ίντα, ο David Martin των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Πρώτα ένα σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με τη μελέτη που μας παρουσίασαν οι δύο επιτροπή. Είναι σαφέ, όπω είπε και ο Παύλο, ότι είμαστε μεγαλύτερε εξαγωγέ ε, γεωργικών προϊόντων στον κόσμο. Οπότε, οποιαδήποτε άνοιγμα των αγορών ε, θα είναι προ όφελο μα. Αλλά όταν εφαρμοστεί η ΣΕΤΑ, για παράδειγμα, ο γαλακτοκομικός μας κλάδος έχει τεράστιες ευκαιρίες εξαγωγής προϊόντων προς τον Καναδά. Έχω δύο ερωτήσεις. Μερικές φορές μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι εμπορικοί μας εταίροι μερικές φορές ε, δεν επωφελούνται δεόντως. Με το Βιετνάμ, για παράδειγμα, έχουμε μία διάταξη ε, ότι οι δεσμοί στο ίνο και ε, ίνο θα κατεβούν στο 0 από 40%. Βέβαια, εξαιτία του ειδικού φόρου κατανάλωση που έχει το Βιετνάμ, ουσιαστικά κυρώνει αυτή την μείωση. Το ίδιο με την Κορέα. Μειώθηκαν οι δεσμοί για το ουίσκι και είναι εύκολη πρόσβαση στις αγορές, αλλά με τις αλλαγές που γίνονται στις τελωνιακές διαδικασίες, τις διαδικασίες εκτελωνισμού ε, εξουδετερώνονται όλα τα πλέον πλεονεκτήματα. Ε, και μία και μόνο εταιρεία έχει, πρέπει να πληρώσει ένα ε, λογαριασμό 5 εκατομμύρια pound τελωνιακούς ε, τελωνιακά τέλη εξαιτία τη αλλαγή τη διαδικασία. Προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι φραγμοί. Εκ μέρου τη ECR από την Επιτροπή Γεωργία, ο κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με ευκαιρία και εγώ να ευχαριστήσω του δύο επιτρόπου και να του καλωσορίσω και να τους ευχαριστήσω για τη δημοσίευση της έκθεσης. Χαιρετίζουμε την έκθεση και βλέπω ότι θεωρούν ότι είναι θετικές οι εμπορικές συμφωνίες για πολλούς κλάδους και μάλιστα βέβαια και σε μερικούς δεν είναι τόσο ευμενείς οι συνέπειες όπως στον τομέα του κρέατος. Και μόνο με τη Μερκοσούρ απειλεί να εξαλείψει την βιομηχανία παραγωγής βόλου κρέατος στην Ευρώπη. Δεν είναι για όλους τους κλάδους λοιπόν ρόδινα τα πράγματα. Και το γεγονός ότι για μερικούς κλάδους είναι θετικά το αποτελέσμα των εμπορικών συμφωνιών δεν είναι δικαιολογία να εφαρμόσουμε την συμφωνία αυτή που θα πλήξει άλλους κλάδους. Επίσης, άλλη επίκριση για την μελέτη. Επικεντρώνοντας μόνο την προσοχή σε οικονομικέ συνέπειες, αγνοούμε τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ωφέλη ή μειονεκτήματα στις αγροτικές περιοχές. Σε πολλές περιοχές ε, της Ευρώπης η γεωργία είναι ε, ο βασικός ε, σύνδεσμος του κοινωνικού ιστού, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως σας ανέφερα του Βόλου Κρέατος. Εγώ πιστεύω ότι η μειονεκτηματα στις αγροτικες περιοχες σε πολλες περιοχες της ευρωπης η γεωργια ειναι ο βασικος συνδεσμος του κοινωνικου ιστου ιδιαιτερα σε κλαδους οπως σας ανεφερα του Βόλιο κρεατος εγω πιστευω οτι η γεωργια θα είναι το αγκάθι των διαπραγματεύσεων, των εμπορικών διαπραγματεύσεων σε πολλές μελλοντικέ συμφωνίες και τώρα που μάλλον παραμερίστηκε η TTIP θα διακοπούν τελικά οι σχετικές διαπραγματεύσει για την TTIP. Άλντε, Γιάννη Χόλντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους για την ισχυρή υποστήριξη της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Ακούτε ε, ποιο είναι το συμφέρον του ελεύθερου εμπορίου για την Ευρώπη. Νομίζω ότι όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, διότι υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός ως προς το ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο γενικότερα να κοιτάξουμε λίγο τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΤΑ. Ήταν οι πιο ανοιχτέ διαπραγματεύσεις που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας όσον αφορά στους καταναλωτές και την προστασία του περιβάλλοντος από την ευρωπαϊκή πλευρά είχαμε το πιο καλό αποτέλεσμα που έχουμε δει ποτέ. Όμως πολλοί πολίτες αντέδρασαν με σκεπτικισμό. Επίσης ε, στις, ε, μετά τις εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε ότι θα έχουμε πρόβλημα και τι θα γίνει και με τη Γαλλία όσον αφορά τις συμφωνίες με και τις νέες εκλογές. Η Κομισιόν έχει μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι το ελεύθερο εμπόριο γίνεται μία βρώμικη λέξη πια, μία λέξη που ακούγεται σαν βρισιά πλέον για τους πολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνη Σεσάρκα από την Ίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους επιτρόπους. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχουμε τώρα τη δυνατότητα να δούμε τα κοινά σημεία μεταξύ δύο τομέων που είναι πολύ σημαντικοί. Βλέπουμε το ε, αντίκτυπο του εμπορίου σε όλους τους τομείς. Είναι δύσκολο σήμερα να το πιστέψει κανείς, αλλά η εικόνα δεν είναι μόνο μαύρη ή άσπρη. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για μας. Ε, με ενθάρρυνε το γεγονός ότι τα νούμερα των εξαγωγών ε, στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής είναι τόσο ψηλά, ειδικά στο τομέα των γαλακτοκομικών έχουμε δει τι γίνεται με το κρασί, με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι θα είμαστε τυφλοί ε, σε προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, ευαισθησίες όπως ας πούμε αυτά που είπε η κυρία Μάλστρομ. Ελπίζουμε το δικαίωμα για τη ρύθμιση να παραμένει ανέπαφο ε, και να προστατεύονται συγκεκριμένοι τομείς όπως θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον και ανάφερε και ο ε, την ανησυχία που υπάρχει σχετικά με την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμο στο τι σημαίνουν αυτοί οι κανόνες εμπορίου και ποιε είναι οι επιπτώσει. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε μία συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την ε, σχέση μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτή η συνάντηση είναι μια δυνατότητα να δούμε την πλήρη εικόνα, να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο για το κάθε μέτρο και αν χρειάζεται να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα μετριάσουν τα προβλήματα αν υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο όταν μιλάμε για αυτές τις συμφωνίες εμπορίου ή και για την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο εθνικό επίπεδο ότι οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια γνωρίζουν ότι αυτά θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα προσαρμογής. Καλό θα είναι να δούμε και αυτό το θέμα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο του Σόλτσε από την ΚΟΕ για την ΙΝΤΑ. Συγγνώμη, θα μιλήσω εγώ εκ μέρους ε, τους. Θα ήθελα αρχικά όσον αφορά τους συναδέλφου ε, ε, να τους ε, ε, ενημερώσω κάτι με τις συμφορίες αυτές θα ξεκινήσουμε μια, ε, μια μάχη ανταγωνισμού την οποία θα χάσουμε ήμουνα σε μια επιχείρηση ε, πατάτας στην Ολλανδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ε, Ολλανδία βρίσκεται στο Χρόνιγεν και εκεί πρέπει να ανταγωνιστούμε εταιρείε οι οποίες έχουν μεγάλες αναλογίες, χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένα ε, ε, τρόφιμα. Στο Μπράμπαντ επίσης ε, μίλησα με γεωργούς που εκτρέφουν χείρους και αυτοί έχουν να ανταγωνιστούν τα κόστη εξαιτίας του κόστους για ανατροφή των ζώων. Γι' αυτό το λόγο αυτοί αντιτίθενται του ΣΕΤΑ και του TTIP ε, και ε, ε, οι αγρότες στην Ολλανδία είναι κατά αυτών. στο ΜΕΙΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάστηκε μια έρευνα πρόσφατα για το TTIP και την αγορά κρέατος στην Ευρώπη. Το βιβλίο λέγεται Selling of the Farm και λέει ότι οι ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μικρότερες και οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν γίνονται θύματα ε, όπως επίσης και ο καταναλωτές και η ε, φύση. Ε, γνωρίζετε αυτή την έρευνα και τι έχετε να πείτε για αυτό. Για την Άγρι, έχουμε τη Μαρία Λίδια Σέντρα Ροντρίγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούω την Επίτροπο Μάλστρομ και τον Επίτροπο Χόγκαν και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Φαίνεται ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Εσείς ζείτε στον κόσμο με τους καρχαρίες, με, τους, με τις πολυεθνικές, με την αγορεπιστιστική βιομηχανία και τους εξαγωγείς. Μόνο λεφτά βλέπετε. Εγώ ζω με τους αγρότες και τις αγρότησες που εξαιτία των δικών σα εμπορικών πολιτικών και τη δική σα ε, κοινή γεωργική πολιτική και των ρυθμιστικών σα πολιτικών, οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τι δουλειέ του και βρίσκονται σε όλο και πιο ευάλωτη θέση. Και όταν μου λέτε ότι θα δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, κάντε πρώτα έναν απολογισμό και πείτε μα πόσε θέσει απασχόληση θα χάσουμε πριν δημιουργηθούν αυτέ που υπόσχεστε, γιατί ε, οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που απορριθμίζουν τα πάντα για να διευκολύνουν χαμηλέ τιμέ για του εξαγωγεί ε, και καλέ συμφωνίε θετικέ για του εξαγωγεί, αυτέ οι συμφωνίε που ανενδίαστα και ανερυθρίαστα καταπατούν όλου του υγειονομικού και περιβαλλοντικού κανόνε, στρέφονται κατά των ε, αγροτών και αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται κατά του ευρωπαϊκού πληθυσμού και στρέφονται και κατά των αγροτών των χωρών εταίρων. Ελπίζω, όπως οι ε, αγώνες των αγροτών σταμάτησαν πολλές εμπορικές συμφωνίες στη Λατινική Αμερική, να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί μην βλέπετε τις εμπορικές συμφωνίες ως πανάκια και αλλάξτε επιτέλους την πολιτική σας. Εκ μέρους των Πρασίνων και από την Επιτροπή Γεωργίας, ο κύριος Μποβέ. Κύριε Επιτροπέ, κύριε Επιτροπέ. Ε, από την αρχή έχουμε πρόβλημα. Άλλο εμπόριο και άλλο ελεύθερες συναλλαγές. Και με βάση αυτό το διαχωρισμό θα πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Επειδή δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω το πρώτο θέμα, να μιλήσω για τη γεωργία. Σήμερα μιλούμε για τον απολογισμό. Αν δούμε ε, τι γίνεται με την παραγωγή χείριου και βόλου κρέατος, Μόνο και με την ΣΕΤΑ με τον Καναδά χάνουμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Αν προσθέσουμε και τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν προσθέσουμε και τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, θα έχουμε πραγματική κρίση της κτηνοτροφίας. Και ποιοι θα είναι ανταγωνιστέ, μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές όπως η Smithfield, που έχουν θηγατρική στον Καναδά την έδρα τους ε, στην ΗΠΑ και οι ιδιοκτήτες είναι Κινέζοι. Αυτό είναι το ελεύθερο εμπόριο. Επίσης, μιλήσατε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οφείλω να σας πω ότι όταν προστατεύουμε 140 γεωγραφικές ενδείξεις από τις 1400, 10% μόνο των γεωγραφικών ενδείξεων προστατεύουμε. Και σήμερα ε, δημιουργήσατε διακριτική μεταχείριση μεταξύ των ε, ονομασιών προέλευσης. Κάνετε διάκριση μεταξύ των ε, ε, προστατευμένων και των μη προστατευμένων ονομασιών προέλευσης. Είναι αθέμητος και παράνομος αυτός ο διαχωρισμός που κάνατε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και για τους Καναδούς αλλά και για τους Ευρωπαίους παραγούς είναι απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες. Η κυρία Μπεγκίν από την EFDD. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ τους επιτρόπους που ήρθαν σε αυτή την επιτροπή εντάχει και εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις αφού έχω την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσω πλήρως. Πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες σίγουρα είναι χρήσιμες συμφωνίες για πάρα πολλούς από τους παραγωγούς μας, αλλά όχι για όλους. Οπότε για να αποφύγουμε να αυξήσουμε τις διαφορές και τις ανισότητες που στοιχώς υπάρχουν στην ε, Ευρώπη μεταξύ, χωρών, μεταξύ των παραγωγών και χωρών, θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι το θέμα του ρυζιού. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις σχετικά με αυτά που κάνει για να περιορίσει τις αγωγείς κυρίως από τι ε, ειδικές ποικιλίε. Κάτι άλλο που αφορά τις κυρώσεις επί της Ρωσίας, αν σε κάποιο βαθμό εργάζεστε, ούτω ώστε να αρθεί το εμπάργκο που ήταν επιζήμιο πάρα πολύ για του παραγωγού όσον αφορά τα γενικά προϊόντα και το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων κάτι που εφήγει από κάποιους ε, συναδέλφους και εγώ πιστεύω ότι δεν αρκούν αυτά που πετύχαμε στον αφορά τη ΣΕΤΑ και αντίθετα η συνάδελφο Ντεκάστρο ρωτά το άλλο και στις άλλες συμφωνίες να φτάσουμε σε αυτού του είδους την προστασία μήπως κινδυνεύουμε ε, να, να χάσουμε τη θέση μας προς ικανοποίηση των άλλων που είναι αντίθετη και άλλο για τις γραφικές ενδείξεις. Τι θα κάνετε. Δεν διαχειρίζονται τα Μήτρο από την Υπηρεσία για την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων της Γενική Γενικής Διευθύνσεως ε, Γεωργίας. Ευχαριστώ. EFTD, John Stuart Agnew. Καλησπέρα, Επίτροποι. Θα μιλήσω για πρωτεΐνες, διότι αφορά τι αρμοδιότητες Εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 30 εκατομμύρια τόνους εισαγωμένων ε, σόγια γενετικά τροποποιημένης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έριξε τον παλάκι στα κράτη-μέλη. Ε, κατά πόσο, να δει κατά πόσο οι καλλιεργητές θα μπορούσαν σε κάτι μέλη να καλλιεργήσουν τη γενετικά τροποποιημένη ε, σόγια. Είπαν όχι τα κάτι μέλη. Μεγάλη υποκρισία αυτή. Πόσο βιώσιμη είναι αυτή η στάση. Να, να προσθέσουμε και άλλες απαγορεύσεις που αφορά το έλαιο κράμβης. Μετά έχουμε τις ζωοτροφές που πηγαίνουν πρωτεΐνες και έχουν λιγότερα εισόδα από την ε, κράμβη, έλαιο κράμβης. Μπορείτε να πείτε μπορεί να χρησιμοποιήσουν φασόλια για τις ζωοτροφές. Μπορεί να μεγαλώσουν μόνο μία πέντε φορές, κάθε πέντε χρόνια με έξι χρόνια. Η σόγια είναι κάθε τρία χρόνια ε, και δεν είναι ποιοτική πρωτεΐνα. Η Κίνα έχει μπει στην αγορά της σόγιας. Άρα μειώνεται η δική μας πρόσβαση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανοιχτά καύσιμα να στεγνώσουμε τη σόγια. Και αν πάρουμε και άλλη απαγόρευση για τα παρασιτοκτόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να καλλιεργούμε τη σόγια. Οι πράσινοι τώρα θα πείσουν τις παγκόσμιες αρχές να μειώσουν την παραγωγή σόγιας στη Λατινική Αμερική για να αντιμετωπίσουν τάχα μου την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα πρόβλημα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Για το ΕΝΕΦ, ο Φιλίπ Λουαζό έχει τον λόγο. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αυτό που αποκαλείται ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι συμφωνίες ε, έντονης απορρίθμισης. Έχουμε διαφορετικά μοντέλα και ως προς το κόστος, ε, τις μεθόδους και τους κανόνες και ενθαρρύνουν μόνο την επαναβιομηχάνηση της γεωργίας. Ε, και Μα υπόσχεστε τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόληση. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να εξακριβώσουμε κάτι τέτοιο. Μάλλον είναι προπαγανδιστικά αυτά τα σχόλια. Γιατί στο μεταξύ πόσε χιλιάδε θέσει θα χάσουμε εργασία, πόσε εκμεταλλεύσει θα, θα βάλουν λουκέτα. Για την ΤΑΦΤΑ, μια αμερικανική μελέτη το 2014 μιλούσε για 600.000 θέσει απόλυτα θέσεων απασχόληση και 50.000 θέσει χαμένε στη Γαλλία. Ε, και μάλιστα θα οδηγήσουν αυτές οι συμφωνίες στο χαμό των λαών μας ενώ θα αυξάνουν τα κέρδη των ε, πολυεθνικών. Είπατε ότι θα είναι κάποιες θετικές συνέπειες. Ποιες ε, για το βόλιο κρέας, ε, απειλές, επίσης υποβάθμιση των προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων και με τον αφεβήτο τρόπο θα κατακλειστούμε από βορειοαμερικανικά προϊόντα που θα είναι πιο φτηνά και που θα παράγονται με πολύ πιο χαλαρές διατάξεις ως προς, την ποιότητα και έτσι θα χάσουμε την αριστεία που είχαμε στα γεωργικά μας προϊόντα με βάση αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Για να μην μιλήσουμε για το ρωσικό εμπάργο που θα οδηγήσει στην αυτοκτονία πολλών ε, γεωργών. Πώς θα διορθώσουμε αυτές τις ε, ανεπανόρθωτες ε, ζημίες πριν να λάβουν χώρα. Από την ΕΝΕΦ, e ο Εντουάρ Φεράν. Μας ε, προβληματίζει το χρονοδιάγραμμα για τη ΣΕΤΑ. Φαίνεται ότι η βιασύνη αυτή κρύβει κάποια προβλήματα. Έχω ερωτήσεις. Ο Καναδά πρόσφατα υιοθέτησε ένα πρόγραμμα ε, χρηματοπιστωτικής βοήθειας 300 ε, εκατομμύριων δολαρίων για τη γαλακτοκομική βιομηχανία. Ε, προβλέπεται αντίστοιχη ενίσχυση για τη δική μας βιομηχανία κρέατος. Επίσης, ε, τι γνώμη έχετε για τις μελέτες που μιλούν ε, για την απώλεια 50.000 θέσεων απασχόληση μόνο στη Γαλλία μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Τρίτον, ε, για τις ονομασίες προέλευσης. Δεν είναι περιθωριακό θέμα. Είναι κέριο ζήτημα αυτό των ονομασιών προέλευσης, γιατί έτσι αναδεικνύεται η αριστεία του ευρωπαϊκού εδάφους. Θα τη θυσιάσετε στο βωμό των ελεύθερων συναλλαγών. Ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στους επιτρόπους για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των συντονιστών. Το πολύ 10 λεπτά ο καθένας. Με την αντίστροφη σειρά από τις αρχές θα ξεκινήσουμε από τον Επίτροπο Χόβιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ο κύριος Βαλές ανέφερε το θέμα της Ουκρανίας. Η συμφωνία με την ε, ε, Ουκρανία είναι στη μελέτη, είναι στη γραμμή βάσης. Είναι ε, στην ουσία μια βάση για όλες τις συμφωνίες που ήδη εφαρμόζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Χρειάστηκε λοιπόν να έχουμε μια απλούστευση για να γίνει καλύτερη η ανάλυση. Η Ουκρανία λοιπόν είναι στην έκθεση και συμφωνώ ότι η σωστή ανάλυση για τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν έχουμε ένα μοντέλο που μας δίνει ακριβώς ε, τη σωστή ανάλυση, οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις ε, απόψεις σας. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ντέσο ότι χρειαζόμαστε ίσους όρους σε επίπεδο εμπορίου. Ο κύριος Μάρτιν ανέφερε το Βιετνάμ και τον φόρο κατανάλωσης ε, που στην ουσία θα δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τα κέρδη που θα έχουμε. Ήμουν στο Βιετνάμ πρόσφατα και συζητήσαμε αυτό το θέμα, το εξετάσαμε με τις βιετναμέζικες αρχές και είδαμε τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιο κυρίαρχο κράτος μέλος τι μπορεί να κάνει με τη φορολογία του, ούτε καν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέσαμε αυτό το θέμα. Ο κύριος ε, Ντεπρές επίσης είπε ότι υποστηρίζουμε το θέμα αυτό ε, γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμφωνώ μαζί του. Κύριε Νίκολσον, να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα του Βοΐου και της Μερκοσούρα έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Θα είδατε ότι ε, στην δεν έχουμε ε, υποκύψεις της φιλοδοξίας ε, των εταίρων μας από τη Μερκοσούρ γιατί ε, υπάρχει το θέμα του βοήου. Και όπως είπε και η κυρία Μάλστρομ, σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο TTIP έχουν μπει όλα αυτά στο ψυγείο. Μάλιστα έχει, πει το θέμα, έχει πάει το θέμα στο δικαστήριο σχετικά με το τι θα γίνει στο μέλλον. Κατανοώ τον σκεπτικισμό και τις ανησυχίες που ανέφερε ο κ. Ρόντεν, όμως το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζονται σωστές και ε, ε, ε, πληροφορίες. Αν δεν είναι πλήρες και ακριβείς οι πληροφορίες σχετικά με το τι περιλαμβάνεται μια, σε μια συμφωνία ελευθερών εμπορίου, θα υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτό που επικρίνει ο κόσμος είναι αυτά που δεν υπάρχουν στις συμφωνίες και είναι Πολύ άσχημα να υπάρχει παραπληροφόρηση στα κράτη-μέλη και οπουδήποτε αλλού. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν ακριβείς αληθείς πληροφορίες που θα μπορούν να πληροφορήσουν τον κόσμο σωστά. Η κυρία ε, Σάκη ανέφερε ε, τα μέτρα για την προσαρμογή που θα πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις. Φυσικά όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και το γνωρίζουν τα κράτη-μέλη, το έχουν ε, στην χώρια πολιτική τους, δεν θα τους το πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ όμως ότι αυτή πρέπει να κάνουν κάποιε τέτοιε προσαρμογές στα πλαίσια της παγκοσμιοποίηση. Επίσης, αναφέρατε το θέμα των καταναλωτών και των παραγωγών. Εγώ θέλω ε, και τους δύο να φροντίσω σε επίπεδο επισητιστικής ασφάλειας, ποιότητας των τροφίμων, και ε, καταλαβαίνετε ότι και οι καταναλωτές αλλά και οι αγρότες πρέπει να παράγουν βιώσιμα έτσι ώστε να έχουμε σωστές αγορές στο μέλλον. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και θα δείτε ότι έχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο χνηλασιμότητας και επιστημιστικής ασφαλείας στον κόσμο. Ίσως να μην ε, συμφωνείτε αλλά σχετικά με όλους τους άλλους είμαστε στην κορυφή. Ε, κυρία Νίσεν, ε, ό,τι και να σας πω σε σχέση με το εμπόριο δεν θα συμφωνήσετε. Ίσως δεν πρέπει να απαντήσω καν στην δήλωσή σας, όμως έχουμε 50 με 60 δις που δίνονται στους γεωργούς κάθε χρόνο, όχι μόνο σε μία φορά, συνεχώς. Και καλό θα ήταν ε, τον Γενάρη του 2017 να ξεκινήσετε να ενημερώνετε τον κόσμο ότι μπορεί να λάβει μέρος σε μία δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα. Πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός ότι ε, δεν δίνεται σημασία σε αυτή την υποστήριξη εισοδήματος στους ε, γεωργούς. Δίνεται ε, αποσυνδεδεμένη βοήθεια στους γεωργούς. Ε, σε πολλές περιπτώσεις το κράτος μέλος είναι αυτό που λαμβάνει την απόφαση και όχι το Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν. Και αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση για τις FTAs και στην Νότια Αμερική, για παράδειγμα. Πρέπει, ας πούμε, σε χώρες όπως το Περού, ο η Κολομβία, η Χιλή, ε, που ε, διαπραγματεύονται μαζί μας να ε, τα γνωρίζουν αυτά. Να τα λέτε λοιπόν σε άλλους και όχι σε μένα. Επίσης, έχουμε την έκθεση του κυρίου Ανδρέου στο Κοινοβούλιο ε, σχετικά με τις προκλήσεις στην απασχόληση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα προστατεύσουμε τα ευαίσθητα προϊόντα. Στη χώρα σας ε, το βόη είναι ένα πολύ μεγάλο ε, προϊόν και αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Βλέπουμε πώς θα προστατεύσουμε με τι μέσα θα προσπιστούμε την ευαισθησία αυτού του προϊόντος στις θέσεις εργασίας. Θα έχουμε πρόβλημα ε, και θα χάσουμε θέσει εργασία. αν ε, συμφωνήσουμε σε όλα όσα μα ζητούν οι Ηνωμένε Πολιτείες. Φυσικά δεν θα συμφωνήσουμε και χρειάζονται δύο για να γίνει μια συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε. Όταν υπάρχουν εξωφρενικές απαιτήσει δεν πρέπει να υποκύψουμε, δεν θα το κάνουμε. Ε, υπάρχουν ας πούμε θέματα που ήταν πολύ ξένα και προς την αγορά του Καναδά και στην ΗΠΑ όπως ήταν οι γεωγραφικές ενδείξεις και ε, κάναμε μεγάλες διαπραγματεύσεις και τώρα έχουμε ικανοποιηθεί ως προς την κάλυψη. Ήταν μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που είχαμε στην αρχή που δεν αναγνωριζόταν τίποτα. Κυρία ο που αντιμετωπίζουμε τη μείωση των ε, εισαγωγών μέσω των δασμολογικών ε, προσωστώσεων. Έτσι το κάνουμε, με αυτό το σύστημα που έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό. Από τότε που έγινα επίτροπος, ε, βγήκα από το γραφείο μου και πήγα στην αγορά για να δω ποια είναι τα γεωργικά προϊόντα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μετά από το ρωσικό εμπάργο. Ε, να δούμε τις επιπλέον ε, προμήθειες που έχουμε για πολλά βασικά προϊόντα. 95% των εξαγωγών που πήγαιναν στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία τώρα ε, πάει στην Άπο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Άρα κάναμε σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια αντικαθιστώντας αυτές τις αγορές φυσικά. Δεν έχουμε την ίδια αξία που θα θέλαμε σε αυτό το στάδιο, αλλά θα προχωρήσουμε, θα μείνουμε πιστοί στα πρότυπά μας και σίγουρα θα μπορέσουμε να ε, επωφεληθούμε από την αυξανόμενο πληθυσμό στην Απανατολή και από την σχέση μας με αυτούς. Τα 30 εκατομμύρια τόνοι που αναφέρατε είναι φυσικά έλλειμμα. Ε, έχουμε συζητήσει για τον κανόνα τρικρόπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για κάποιες ε, προς των γεωργών. Το είπαμε στους γεωργούς, αλλά αυτοί ε, δεν επέλεξαν τα ε, προϊόντα που εμείς τους υποδείξαμε, αλλά άλλα. Άρα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ε, σε πρωτεϊνούχα φυτά, σε φασόλια και αντίστοιχα προϊόντα και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε έλλειμμα, πρέπει να εισάγουμε από διάφορα μέρη του κόσμου και θα δείτε ότι υπάρχει και ανησυχία στην κοινωνία που αντικατοπτρίζεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και για την έγκριση των αδειών παραγωγών. Ε, επειδή μπορεί να επωφελούνται οι ανταγωνιστές. Ο κύριος Λεζούρ και ο, ο κύριος Φεράν ανέφεραν θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση. και την υποστήριξη για το βόλιο κρέας. Όπως ξέρετε, Υποστηρίζουμε την βιώσιμη παραγωγή βοήου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τονίζω τη λέξη βιωσιμότητα γιατί η αγορά, εντάξει, είναι δικαίωμα των παραγωγών να παράγουν προϊόντα, αλλά ε, είναι και το σωστό που πρέπει να γίνεται και για την αγορά να υπάρχει βιωσιμότητα. Τώρα για τις ε, θέσεις εργασίας που θα χαθούν, τα τελευταία νούμερα να γνωρίζουν ε, ότι θα υπάρξει μείωση του αριθμού των ανθρώπων στην ε, πρωτογενή παραγωγή, αλλά θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ε, σε άλλους τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 44 εκατομμύρια άτομα στη Γεωργία συνολικά και θα μειωθούν αυτοί που βρίσκονται στο πρωτογενή τομέα και γιατί συνταξιοδοτούνται και γιατί υπάρχουν πολλές ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, λόγω εξορθολογισμού, αλλά θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ε, στους τομείς προστιθέμενης αξίας. Ευχαριστώ. Τέλεια και ιδίω όσον αφορά το χρόνο. Η Επίτροπο, η κυρία με έχει τα λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Απάντησε κάποιε ερωτήσει ο Επίτροπο Χόγκαν. Θα επί των άλλων. Βέβαια, ο αντίκτυπο όσον αφορά τα φυτογενομικά στι εμπορικέ συμφωνίε είναι πολύ σημαντικό. Όπω ο Επίτροπο ε, Χόγκαν δεν υπάρχει άριστη μέθοδο. Μπορούμε να συνεργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Επίτροπο Αντροκάητη για να βελτιώσουμε την όλη ανάλυση μα για τα μεγαλύτερα προβλήματα, τόσο ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στι εμπορικέ συμφωνίε αλλά και στην γενική προσπάθειά μα να απευθυνθούμε σε τρίτε χώρε. Ισότιμε συνθήκε. Για να δημιουργηθεί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά να απαγορεύεται. Δηλαδή, το βόλιο κρέας που έχει, το έχουν επεξεργαστεί ε, με ορμόνες απαγορεύεται. Δεν μπορεί να απολυθεί τέτοιο βόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία και παύλα. Και υπάρχει νόμος περί Τα τρίτα μέρη θα πρέπει να συμμορφωθούν. Έχουμε νόμους για την ευημερία των ζώων όσον αφορά τη σφαγή και μεταφορά και συμμόρφωση με αυτούς τους νόμους είναι υποχρεωτική για τα τρίτα μέρη. Διεξάγουμε ελέγχους λοιπόν και άλλοι κανόνες για την ευημερία των ζώων υπάρχουν που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη στι διάφορε διεθνείς συζητήσει και στο Διεθνή Φορέα για την Επιμερία των Ζώων και στη ΣΕΤΑ δημιουργήσαμε ομάδα εργασία για την Επιμερία των Ζώων για να επεξεργαστούμε από κοινού τα θέματα. Όσον αφορά τι γεωγραφικέ ενδείξει, να προσθέσω σε αυτά που έλεγε ο Πίτροπο Χόγκαν. Έχουμε την προστασία περίπου 1.400 ονομασιών στην Ευρώπη. Αυτό παραμένει στι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε. Τα κράτη-μέλη μα δίνουν ένα κατάλογο με τι σημαντικότερε ενδείξει προέλευση για εξαγωγή σε αυτέ τι χώρες. Πολλές γεωγραφικέ ενδείξεις προστατεύονται εδώ, αλλά δεν εξάγονται σε αυτή την άλλη χώρα. Κάνουμε έναν κατάλογο λοιπόν με τα... τις που έχουν προτεραιότητα και πετύχαμε 140, 160, 170 με κάποιε χώρε και είναι επίτευγμα. Πολλές άλλες χώρες δεν το έκαναν αυτό πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύονται τα άλλα προϊόντα. Όσον αφορά το, το και την Κορέα, είμαστε σε επαφή με τους Κορεάτες για το TTIP επέστρεψα τη ΣΥΠΑ σήμερα το πρωί και συζήτησα εκεί με τον πρέσβη τον Κεφόρμαν αποτιμήσαμε το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το τέλος του έτους θα κάνουμε μια αποτίμηση να δούμε μετά τρία έτη διαπραγματεύσεων που βρισκόμαστε θα υπάρξει κάποια παύση, μεγαλύτερη παύση πιθανότατα στη διαπραγματεύση TTIP με τη νέα κυβέρνηση ξέρουμε ελάχιστα όσον αφορά τις προτεραιότητες του Πρόεδρου Τραμπ Ποτέ δεν ανέφερε το TTIP. Uh, Και για την ώρα θα παγώσουν οι διαπραγματεύσει. Πώ θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη για τη συμφωνίε ελευθερού ε, εμπορίου ήταν η άλλη ερώτηση. Τεράστιο θέμα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εμπορικέ μα συμφωνίε είναι αποτελεσματικέ, αποδοτικέ, ανταποκρίνουν τι ανάγκε των ανθρώπων, δίνουν αποτελέσματα στου καταναλωτέ, μικρομεσαίε επιχειρήσει κλπ. κλπ ότι πραγματοποιούνται διαφανώς, προθούμε και πολύ μάλιστα τη διαφάνεια, το Συμβούλιο αρνείται να δημοσιεύει κάποιες εντολές. Σας ενθαρρύνω να πιέσετε το Συμβούλιο από αυτού μαζί μας και θα εξακολουθούμε να είμαστε στο μέτρο του δυνατού διαφανής και να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εμπορικές μας συμφωνίες συμπεριλεύουν κάποιες, κάποια πρότυπα, αξίες, προδιαγραφές, προδιαγραφές και αξίες να προωθούμε από εργασιακά δικαιώματα, ανθρωπίνα δικαιώματα, περιβαλλοντικά πρότυπα, το δικαίωμα ρύθμιση κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να προωθούνται, θα πρέπει να συνομιλούμε τα κράτη-μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια, με την κοινωνία των πολιτών το κάνουμε, αλλά πρέπει να κινηθούμε περισσότερο. Και τα κράτη-μέλη από τη στιγμή που έδωσαν τη συνένεσή του σε μια διαπραγματευτική εντολή και με ομοφωνία δίνουν τη διεντολή μας που διαπραγματευόμεθα θα πρέπει να βγουν και να πάνε στις χώρες τους υπεύθυνοι και να πούν κοιτάξτε συμφωνήσαμε να διαπραγματευτούμε με το Μεξικό. Θα είναι πολύ καλή συμφωνία αυτή. Γι' αυτό και τον τάδε και το δίνω λόγο. Για ακούστε τι ανησυχίε του κόσμου και ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρο, όχι μια εβδομάδα πριν την κύρωση. Διότι τότε αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πιο δραστήριοι. Και εκεί έχουμε αποτύχει όλοι. Δηλαδή να εξηγήσουμε, να συνομιλήσουμε με του πολίτε, να ακούσουμε τι ανησυχίε και να συμπεριλάβουμε τι ανησυχίε, να αισθανθεί ο κόσμο ότι εισακούγεται. Και να εξασφαλίσουμε ότι εκείνοι οι οποίοι χάνουν από την παγκοσμιοποίηση και πολύ σπάνια απόλυε θέσει οφείλονται σε εμπορική συμφωνία οφείλεται η απώλεια εργασίων λόγω παγκοσμιοποίησεως, ε, ε, τεχνολογικής ε, προόδου κλπ. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και οι τιμένοι στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα εργαλεία τόσο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, τόσο ώστε ο κόσμο να έχει πραγματική κατάρτιση, υποδομέ, δεξιότητε για να αλλάξει θέση εργασία. Κάτι πράγματα μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του πόρου μα με ευφιέστερο τρόπο, αλλά τα περισσότερα είναι στα χέρια των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται ο κατάλληλο ε, συντονισμό, καλύτερο συντονισμό. Τέλο, υπάρχουν διάφορε εκθέσει που προσμετρούν τον αντίκτυπο τη TTIP τη ΣΕΤΑ, παραδείγματο χάρη. Περισσότερε εκθέσει και μελέτε δείχνουν την ίδια κατεύθυνση. Αύξηση απασχόληση, αύξηση επενδύσεων, αύξηση ανάπτυξη. Και υπάρχει μια μελέτη που πολλοί από εσά αναφέρατε που γίνεται με εντελώ διαφορετική μεθοδολογία που ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για εμπορικέ συμφωνίε. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τα αποτελέσματα τη ελόγω μελέτη και κανένα ε, σοβαρό ακαδημαϊκό δεν συμφωνεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι εμπορικέ συμφωνίε πάντα οδήγησαν σε θέσει απασχόληση, ανάπτυξη και ανάπτυξη επενδύσει. Είδαμε επιτυχέστατε συμφωνίε. Η συμφωνία με την Κορέα οδήγησε σε 250.000 θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Με τον Επίτροπο Χόγκαν σας δώσαμε ένα παράδειγμα αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων για τον αγροτροφημικό τομέα. Αυτό οδηγεί σε ανάπτυξη και επενδύσεις. Ε, και βέβαια και άλλες συμφωνίες είδαμε κατά το παρελθόν που πάντα οδήγησαν σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ιστορικά αυτές ενδείξεις έχουμε και γι' αυτό ε, εκεί στηριζόμαστε να προβλέψουμε. Δεν θα ωφεληθεί εξίσου κάθε χώρα ούτε κάθε τομέα. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να κάνουν εθνικές προβλέψεις και να προσπαθούν να καλύψουν και να ενημερώσουν τους ευάλωτου τομεί έγκαιρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ σταματώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Χόγκαν θα απαντήσει σε απάντηση τη άλλη. Ευχαριστώ Επίτροπε. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Δίνω την Προεδρία στον Συμπρόεδρο. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχουμε 30 περίπου ομιλητές στο κατάλογο. Ένα λεπτό στο καθένα. Και στο λεπτό πάνω θα σηκώνω το σφυράκι μου. Ο κύριος Τσούλο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, επιτρόπους. Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω ενθουσιώδης ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Δεν είμαι όσο ενθουσιώδης είσαστε εσείς για τα αποτελέσματα στις συνθήκες και συμφωνίες. Για τους ίδιους λόγους που προβάλλατε εσείς δεν είμαι ενθουσιώδης. Το είπε η Επίτροπος η κυρία Μάστροπο. Ε, δεν έχουν τα ίδια ωφέλη οι, όλες οι χώρες και όλοι οι τομείς από αυτές τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίες. Άρα ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων. Και επειδή προσέχουμε τους παραγωγούς και τους πολίτες, και γι' αυτό θέλουμε διαφορετική προσέγγιση. Είπατε ότι οι μελέτες αφορούν μόνο το 30% των, εξαγω... των προϊόντων που εξάγονται. Πού είναι τα άλλα 70% οι μελέτες που καλύπτουν το υπόλοιπο 70% των προϊόντων. Εκεί γίνεται διαφορά. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να συνάπτουμε πάση θυσία τις συμφωνίες, θα πρέπει να βασιστούμε επί των ποιοτικών τομέων που σήμερα δεν καλύπτονται όπως είναι το κρασί, ε, μεταπημένα προϊόντα, το έλαιο και διάφορα προϊόντα που τελικά θα υποβιβαστούν από πρώτη κατηγορία σε δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, μια ερώτηση που στον κύριο Χόγκαν. Μακροπρόθεσμα για τον αγροτροφημικό τομέα, ποιο είναι το ρασμά της Ευρώπης, για την παραγωγή και για την εσωτερική κατανάλωση. Προς τα πού πηγαίνουμε. Ο κύριος Σούλτς. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, επιτέλους έχουμε μια μελέτη, γιατί επανειλημμένο ζήτησα μια μελέτη που να συγκρίνει με οριζόντιο τρόπο όλες τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Βέβαια, άλλα τα συμφέροντα της αγροπιστικής βιομηχανίας και άλλα τα συμφέροντα των γεωργών. Γιατί η αύξηση της εξαγωγής τυριών, για παράδειγμα, δεν ε, θα οδηγήσουν ε, αυτόματα σε αύξηση της τιμής του γάλακτος. Οπότε, το θέμα είναι να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των γεωργών στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και όχι μόνο της αγροπιστικής βιομηχανίας. Ένα από, τα, από τους αρνητικούς τομείς είναι το βόιο, ρύζι, ζάχαρη, ε, πουλερικά. Επίσης ε, έχουμε και το παράδειγμα της συμφωνίας με την Ουκρανία που προϊόντα της Ουκρανίας κυρίως εξάγονται προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ εμείς δεν έχουμε διέξοδο για τους παραγωγούς μας. Μην ξεχνάτε λοιπόν και αυτούς τους παραγωγούς για τους τέσσερις ευαίσθητους τομείς που σας ανέφερα. Η κυρία Ράς. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η μελέτη σας, που είναι θεωρητική, δεν, υπόψη, δεν λαμβάνει υπόψη κάποια μέτρα μηβαίας απελευθέρωσης και τα οικονομικά μέτρα. Για παράδειγμα, η μείωση μη δεσμολογικών φραγμών, όπως είναι των φυτοϊγειονομικών και υγειονομικών μέτρων. Γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια αμοιβαιότητα, ώστε όλα όσα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρούν τις δικές μας προδιαγραφές. Γιατί αν έχουμε περιπτώσεις λοιπούς ελέγχου και ε, ασθένειες όπως η ξυλέλα φαστιδιώσα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω χαλαρότητας και έλλειψης ελέγχου, τι θα κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν οι μελέτες να είναι πιο διεξοδικές, πιο εμπεριστατωμένες. Γιατί είναι κρίμα για τα προκυπευτικά, για το ελαιόλαδο, για τον ίνο, να μην γνωρίζουμε τι δυναμικό και τι ευκαιρίες θα δημιουργούνται για αυτούς τους κλάδους ε, λόγω των συμφωνιών. Η κυρία Ρενά. Ευχαριστώ. Έχω πολλές παρατηρήσεις. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στην Νότιο Κορέα και συμφωνώ κυρία Μάλστρο μαζί σας ότι όντως είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα ε, από τη συμφωνία αυτή, κυρίως όμως για τη χημεία, χημική βιομηχανία, την ενέργεια, τη χρηματοπιστωτικά ε, χάρη στη συμφωνία. Και βέβαια οι εμπορικέ συμφωνίε ευνοούν τι πολυεθνικές και του μεγάλου κλάδου και όχι τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και το είδαμε αυτό στη συμφωνία με την Νότια Κορέα. Ποιοι επωφελήθηκαν. Αφήστε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό έλεγχο, ε, αντίκτυπο της συμφωνία με την Νότια Κορέα. Επίση, ε, πώ επηρεάζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το ύψο των μισθών στην Κορέα. Γιατί είχαμε κάποια πρόοδο για, για τη βιομηχανία, αλλά στους άλλους, στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς είχαμε αντίστοιχη πρόοδο. Επίσης, στην Νότια Κορέα, η, ο βασικός δικαιούχος και αυτός που θα ωφεληθεί περισσότερο από τη συμφωνία είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα έχουμε όμως τον Brexit, ελήφθη υπόψη και τι θα γίνει μετά τον Brexit. Και για τη ΣΕΤΑ, μιλήσαμε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 10% καλύπτονται, με πάρα πολλές εξαιρέσεις. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εξαιρέσεων στις γεωγραφικές ενδείξεις Επίσης, ο έλεγχος ε, του βόλιου κρέατος με ορμόνες. Πολύ φοβάμαι ότι θα ξεσπάσει νέο επιστημιστικό σκάνδαλο στην Ευρώπη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής βόλιου κρέατος. Ο κύριος Αγαπητέ Πρόεδρε, φαίνεται ότι ε, ανοίγουμε το δρόμο σε νέες αγορές, αλλά οι συμφωνίες αυτές αποτελούν μεν έναν καλό τρόπο λειτουργίας, αλλά η Γεωργία θεωρεί ότι αποτελεί το αντάλλαγμα. Σας ευχαριστώ για το είναι έκθεση επιπτώσεων. Είναι μια έκθεση η οποία αγνοεί όμως τις αγορές, ε, τα συμβάσεις που ήδη έχουν συναυθεί και θα πρέπει να προσθέσουμε αυτές τις συμβάσεις αυτές που προβλέπονται και να γνωρίζουμε ακριβώς τον αντίκτυπο στον τομέα. Όσον αφορά του αριθμού για το κρέα, με εξέπληξαν τα αποτελέσματα γιατί είναι πολύ ε, κάτω από τα σύνολα που εγώ είχα βγάλει. Αν θέλουμε ε, συμφωνία με τη Μερκοσούρ, θα έχουμε έλλειμμα, έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 3,5 περίπου δις ευρώ ε, και δεν θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε τα μέτρα για να αντισταθμίσουμε όλα αυτά τα σημεία στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ε, για το κρέας. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο οι εμπορικές συμφωνίες ε, γενικότερα ήταν ε, θετικές για την γεωργία, όπως είναι για παράδειγμα τα χαλοκτοκομικά, αλλά και το χοιρινό κρέας, το βόλιο όμως αποτελεί πρόβλημα και λαμβάνοντας υπόψη αυτά, ε, στην ε, περίπτωση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής θα υπάρξει κάποια υποστήριξη για το βόλιο ή θα υπάρξουν κάποια κίνητρα προς τους αγρότες ούτως ώστε να υπάρχει μια ποικιλία μεταξύ των διαφόρων ειδών γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω την συνέπεια, για, για τις συνέπειες των ρωσικών απαγορεύσεων. Ως μέλος της αποστολής ε, ε, ΑΣΕΑΝ επισκέφθηκα ε, προσφάτως την Ινδονησία και εκεί είδαμε τις εξελίξεις. Ο κύριος Ταραμπέλα. Κυρία Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Ας μιλήσουμε για τη μελέτη σας, που παρουσιάζει ένα σενάριο δύσκολο για, παραγωγή, για κλάδους όπως ο ρύζι, ζάχαρη, πουλερικά, βόλιο. Εκεί και οι τιμές μειώνονται και η παραγωγή. Αυτό ήταν το συντηρητικό σενάριο. Ε, επίσης, για το γάλα μας υπόσχεστε λαγούς με πετραχίλια. Ε, δεν νομίζω. Ε, λαμβάνει το σενάριο την πιθανότητα αύξηση τη τιμή 2 με 7%. 25 λεπτά το λίτρο είναι αυτή τη στιγμή ε, η, η, τιμή του γάλακτος και με την πρόταση που κάνετε άντε να γίνει 26-27, ελάχιστη τιμή. Οπότε πλάνει το θετικό σενάριο. Υπερβολικά ε, φιλελεύθερη είναι η προσέγγιση της κυρία Μάρστρομ και τα, πλεονεκτήματα θα είναι τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για μερικούς οικονομικούς κλάδους και τη γεωργία. Επίσης, ε, ε, στην αγορά του Ντακάρ εξάγουμε το πλεόνασμα γιατί καταργήθηκαν οι μηχανισμοί ρύθμισης με, με αποτέλεσμα η, ο ανταγωνισμός είναι ακόμη χειρότερος με τους αφρικανούς μικροκαλλιεργητές μετά τη συμφωνία. Ε, εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι όλες οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ε, αυξάνουν την ευημερία των πληθυσμών που υποφελούνται από τέτοιες ε, συμφωνίες. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπω ότι η σωρευτική επίπτωση είναι υψής της σημασίας για την μακροπρόθεσμη εμπορική πολιτική. Ε, πολλά από τα ερωτήματα τα οποία είχα ε, τέθηκαν ήδη, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επαναλάβω τα συγκεκριμένα ερωτήματα όπως είναι για την αντιμικροβιακή αντίσταση. Κύριε Μαγκίνες, Ευχαριστώ Πρόεδρο, Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ και τους ε, επιτρόπους. Όσον αφορά το τελευταίο σχόλιο, η αναφορά αυτή επιβεβαίωσε για το ότι ανησυχούμε συγκεκριμένα για το ε, βόλιο κρέας και τι, πώς θα το λάβει υπόψη της Κομισιόν αυτό, διότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα κάνουμε γνωρίζοντας όλα αυτά, Κυρία Μάνστροβ, είπατε ότι υπάρχουν ελλείμματα στην όλη ανάλυση, όμως από τη δική μου πλευρά είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό, τουλάχιστον αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα, όμως ανησυχώ και ε, ενδιαφέρομαι να μάθω τις ε, συνέπειες. Μιλήσατε επίσης για το ελεύθερο ε, εμπόριο. Όμως ο κύριος Γιούγκερ δεν είπε για δίκαιο εμπόριο, όχι μονάχα για ελεύθερο εμπόριο. Οπότε μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τις λέξεις αυτές. Και τέλο υπάρχει συζήτηση σχετικά με μηχανισμούς Άμυνα εμπορίου σε όλου του τομεί. σε περίπτωση που η αγορά δεν λειτουργεί καλά, τότε θα έχουμε μέσα για να επέμβουμε. Θα το έχουμε αυτό ε, σε τι μορφή. Κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο θέματα που δεν τα θίξατε. Θα τα θέσω εγώ πολύ συγκεκριμένα. Οι ερωτήσει μου απευθύνονται προς τον Επίτροπο Χόγκαν, είναι της δικής του αρμοδιότητας. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, σε ό,τι αφορά την επιστηστική ασφάλεια, την υγεία και την αρχή της προφύλαξης, που την εφαρμόζουμε μερικές φορές με ακραίο τρόπο, οδηγούν στην εξάλληψη πολλών δραστικών ουσιών που αποτελούν που περιέχονται στη σύσταση των φυτογενειομικών προϊόντων. Έχουμε αφαίρεση τέτοιων δραστικών ουσιών με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες οι γεωργοί, για να μην μιλήσουμε για το κόστος. Επίσης, με την γονιδιακή τεχνολογία, είδαμε τι προβλήματα έχουμε με τη γλυφοσάτη και τη μεταζώνη ενώ άλλες χώρες δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Επίσης η μελέτη αναγνωρίζει ότι το ρύζι θα είναι από τα προϊόντα που ε, θα έρθουν σε, δυσκο... σε δυσμενή θέση με, την... Ε, με τις εμπορικές συμφωνίες. Γιατί να μην λάβετε υπόψη και τις μεσογειακές καλλιέργειες που είναι το, το καλλιέργειες ε, ελαιοδέντρων, η παραγωγή ελαιολάδων, πορεκυπευτικών και επίσης να φροντίσετε να κάνετε κάτι για το ρύζι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε Χόγκαν, Αναφερθήκατε στην πολιτική φύση του εμπορίου που είναι πολύ έντονη. Πουθενά δεν φαίνεται περισσότερο από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ζωτική σημασία για του Ευρωπαίου γεωργού. Στοιχεία τη Eurostat μα λένε ότι το 2014 το Ηνωμένο Βασίλειο εξήγαγε γεωργικά αγαθά που άξιζαν 16 δι προ την Ευρώπη, αλλά εισήγαγε αγροτικά προϊόντα που άξιζαν 40 δι από την Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερο αγωγέα από γαλλικέ ακμεταλλεύσει, 41% που πίνουν ε, στην ε, ε, από την ραντική αγορά πάνε και το Βόιο πάει στην, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και 30% του υγρού γάλακτος από τη Βόρεια Ιρλανδία πηγαίνει στην αγορά της δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ποιοι εγγυήσει μας δίνουν οι δύο επίτροποι σε όλους τους γεωργούς μας ότι θα επιδιώξουν να υπάρχει ε, μια αμοιβαία επωφελής πρόσβαση στην αγορά και για τα δύο διαπραγματευόμενα μέλη. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Όπως και οι προλαλήσαντες η μελέτη φαίνεται ότι καλύπτει τα διάφορα ερωτηματικά των Ευρωπαίων γεωργών που θεωρούν πολύ συχνά ότι αυτή, αυτός ο δρόμος προς συμφωνίες γίνεται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη δραστηριότητά του. Έχω δύο σημαντικά συμπεράσματα ότι η παγκόσμια αυτή συναλλαγή είναι υποφελής αλλά εκθέτει κάποιους, εκθέτει τομές σε περισσότερους κινδύνους. Μια εμπορική συμφωνία είναι μια συμφωνία που επιτρέπει την ισορροπία μεταξύ ανοίγματο μια αγοράς για τις εξαγωγές και τη διαφύλαξη ευαισθητήτων τομέων. Δεύτερο συμπέρασμα. Έχουμε κάποιε επιφυλάξει. Πρέπει ο κάθε τομέα να εξεταστεί. Ο τομέα των απορρικεπιστικών και των λαχανικών ε, που δίνει πολλέ θέσει εργασία και είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη λησμονήθηκε. Έχουμε 7 συμφωνίε, 12 η συμφωνία με το Μαρόκο και αντίκτυπο που έχει τον τομέα τη ντομάτα δεν μελετήθηκε, δυσμονήθηκε. Και ένα στοιχείο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ο αντίκτυπο όσον αφορά τη δική μα των τιμών στη Γεωργία δεν μελετήθηκε. Και αυτό είναι πολύ επιζήμιο. Θεωρεί η μελέτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ομοιογενή οντότητα, οπότε δεν έγινε μελέτη αντικτύπου κατά κράτο μέλο και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Και τέλο, δεν ελήφθησαν υπόψη οι πολιτικέ δημόσια παρέμβαση που εφαρμόζονται από τα υποτευόμενα μέρη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το ίδιο και για τομεί που θα έχουν επηρεαστεί από αυτή τη συμφωνία που σήμερα δεν βρίσκουν στα εργαλεία τη κοινή ερωτική πολιτική κάποια απάντηση. Η κυρία Κάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πολύ σύντομα θέλω να αφαιρθώ στι συνέπειε των εμπορικών συμφωνιών. Είναι καταστροφικέ αυτέ οι συμφωνίε για του ανθρώπου, τα ζώα και το περιβάλλον. Είναι καταστροφικέ για του καταναλωτέ. Επίση, η παραγωγή θα αυξηθεί αλλά ο πλανήτης μας δεν μεγαλώνει παρομοίως. 3,5 εκατομμύρια περιφερειακές κυβερνήσεις έχουμε, ε, έχουμε πολίτες, ζώα, όλοι αυτοί δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο. Και είναι κρίμα που η Επιτροπή Γεωργίας και αυτή δεν παίρνει το ρόλο της στα σοβαρά και μένει εκτός νυμφώνος. Αν γνωρίζετε ποιος είναι αντίκτυπος της ΣΥΤΑ για τον αγροτικό τομέα, Πώς μπορείτε να είστε υπέρ αυτής της συμφωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τους γεωργούς μας. Ο κύριος Μάτο Ντροβέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι αποφελείς, αλλά αυτό είναι, που είναι σίγουρο είναι ότι είναι αναπόφευκτες. Πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι στις συμφωνίες αυτές τα σπασμένα τα πληρώνει πάντα η γεωργία. Και αυτό μας ανησυχεί. Πολλό δε μάλλον ε, στις απόμακρες περιοχές, στις εξόχως απόκεντρες όπως τα Κανάρια νησιά. Εκεί τα προβλήματα επιδεινώνονται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Βέβαια έχουμε κάποιες ρήτρες διασφάλισης, αλλά ξέρετε ότι δεν αρκούν και είναι και αναποτελεσματικές πολλές φορές. Παρακαλώ λοιπόν κάντε μια προσπάθεια ώστε να εκπονήσετε μελέτες επιπτώσεων των συμφωνιών και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές πριν τι υπογράψετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ τους επιτρόπους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των παραγών στη χώρα μου, στη Βουλγαρία. Και ισχύει αυτό που λέω και για τους γεωργούς σε άλλες χώρες. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι νέοι γεωργοί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αύξηση του ανταγωνισμού που θα προκύψει τι συμφωνίες. Η Καναδική Γεωργία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της χώρας του Καναδά και 35 εκατομμύρια πληθυσμό. Και εμείς έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους. Το άνοιγμα της αγοράς μας θα αφελήσει τους δικούς τους γεωργούς. Και οι συνέπειες για τους Ευρωπαίους γεωργούς σίγουρα θα είναι ε, κάτι αρνητικό και αυξάνεται επίση η διαφορά μεταξύ εμπορικών κέντρων και περιφέρεια. Εξαγωγέ λένε, λένε ότι η ΣΕΤΑ θα αυξήσει αυτή την τάση και θα πληρώσουν την ύφη τελικά οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Σύμφωνα με αξιολογήσει ειδικών, χιλιάδε θέσει εργασία θα εξαφανιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω ε, από τον αγροτικό τομέα, αν τελικά ισχύσει υπό την παρούσα μορφή τη η ΣΕΤΑ. Πώς θα πείσουμε τους μικρούς ε, γεωργούς από την περιφέρεια ότι αυτή η συμφωνία είναι επωφελής για αυτούς. Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή είπατε ότι άνθρωποι εκτός της ε, αγροτικής ε, κοινότητας το αγνοούν όμως είναι ντροπή το γεγονός ότι η Επιτροπή ε, Άγρια αποφάσισε να το αγνοήσει και να μην εκφράσει μια θέση για το ΣΥΤΙ. Ο Επίτροπος Χόντογκαν είπε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ε, σωστέ πληροφορίε εκεί έξω. Συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή σχετικά με το πώ διαπραγματεύεστε, διότι δίνοντας στην προσπάθεια να δώσετε αληθινές ε, και ακριβείς πληροφορίε πήγα στο αναγνωστήριο και θα έλεγα ότι ήταν πιο δύσκολο να, να περάσω το τείχος του Βερολίνου παρά να ε, φτάσω αυτές τις πληροφορίες. Εγώ λοιπόν το αποκαλώ ντροπή αυτό, διότι είναι ε, πιο εύκολο να βρούμε ε, απλές πληροφορίες εάν ε, δεν σου επιτρέψουν να έχεις ένα φύλλο χαρτί, φωτογραφίες, να πάρεις φωτογραφίες. Τότε είναι αδύνατο όντως να δώσεις αυτές τις πληροφορίες παρακάτω και σε άλλους. Έτσι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες ε, διότι το θέμα δεν είναι μόνο πώς θα παράγουν περισσότερα αλλά και πώς θα πουλάνε τα προϊόντα τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες παρά τα όσα λένε κάποιοι. Έχουμε 1,5 δις αν κατάλαβα σωστά ε, εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε και αριθμό για τις εισαγωγές που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια κατανομή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά αυτά τα 11,5 δις αυτό το ποσό πώς κατανέμεται σε επίπεδο κρατών μελών ποια είναι η συνεισφορά στις εξαγωγές για κάθε κράτος μέλος, γιατί θα ήθελα να ξέρω αν μόνο τα ε, δυτικά κράτη είναι αυτά που εξάγουν. Ίσως ε, και οι ανατολικές χώρες βέβαια να έχουν κάποια συμμετοχή. Όσον αφορά στην ε, συμφωνία με την Κίνα είπατε ότι μπορούμε να έχουμε 7 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κάποια συμφωνία. Ποιες είναι αυτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ολλανδία είναι χώρα εξαγωγική, εμπορική. Το έχουμε ε, μέσα στην ιστορία μας. Αυτό μας έκανε μια μεγάλη χώρα. Δυστυχώς όμως ε, είμαστε ε, ιδιαίτερα επικριτικοί όσον αφορά στην ΣΕΤΑ και είμαστε σε καλύτερη θέση να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Κύριε Χόγκαν, μιλήσατε για τα βιώσιμα προϊόντα. Η ερώτησή μου είναι, έχουμε το σχέδιο Juncker, ε, απομένουν 500 ή ίσως 400 δις ε, δεν, ακόμα. Δεν θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε για ένα project που θα λύσει τα προβλήματα, γιατί τα βιώσιμα προϊόντα έχουν πολύ ψηλά στάνταρα στην Ευρώπη και σίγουρα στην Ολλανδία. Και αυτό είναι και το ζήτημα, το να επιτύχουμε αυτές τις υψηλές ποιότητες. Ο κόσμος μιλάει για την ναύτα, για τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν ήδη από το 1994 και μετά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ε, ε, γιατί από το 1994 έκλεισαν πολλές εκμεταλλεύσεις και σε άλλες ε, χώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσατε για τα ταξίδια που κάνατε. Είστε πολύ ενεργός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να, ε, να γνωρίζουμε ότι έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους που σας συνόδεψαν και είπαν πολύ καλά πράγματα. Δεν έχω φόβο για την αγορά. Αυτό όμως που με εκπλήσει είναι ότι τώρα κάνουμε μία μελέτη όπου βλέπουμε ακριβώς αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλες επιδόσεις όπως ας πούμε ο ίνος, ένα από τα μεγαλύτερα προϊόντα ή μιλάμε για το βόιο κρέας ή για το σιτάρι. Έχουμε επίσης τα επεξεργασμένα προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για τις ε, ονομασίες προέλευσης ε, Καταλαβαίνω ότι το καλύτερο θα ήταν να τα ε, προστατεύσουμε όλα, αλλά όταν ε, βλέπουμε αυτό το κατάλογο που υπάρχει ήδη, ε, βλέπω ότι πάντοτε το ίδιο νόημα υπάρχει και θα ήθελα να μάθω κατά πόσο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και ε, τους Επιτρόπους. Πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει πάνω σε αυτό και αποτύχαμε. Νομίζω ότι θα ήταν το θέμα ότι η επανένωση ήταν διαφορετική και τα ρωσικά ήταν διαφορετική γλώσσα τότε όσον αφορά την προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα όμως, όμως ε, ε ανησυχώ για ζητήματα όπως είναι τα πρότυπα ε, παραγωγής ε, και διανομής. Σε άλλες εποχές ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε αυτά τα πρότυπα και ίσως να τα βελτιώσουμε κιόλα αν είχαμε ιδέες εξετάζοντας τι άλλο υπάρχει στον κόσμο. Διότι θα μπορούμε να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, Επίτροπε Μάλμστρομ. Ε, σας άκουσα αρκετές περιφορές ε, και μου φάνηκε γνωστό και πρώτη φορά το συνειδητοποίησα. Είστε ο Ντόναλτ Τραμπ της ευρωπαϊκής πολιτικής διότι δεν μπορείτε να ακούσετε τις ανάγκες. Δεν, ακούτε τις ανησυχίες για τις διάφορες συμφωνίες παρόλο που οι αγρότες, οι κοινωνίες των πολιτών, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σας έχουν πει ότι βρίσκεται στη λάθος κατεύθυνση και όπως ο Τραμπ αρνείται να ακούσει τους ειδικού έτσι και εσείς δεν ακούτε αυτές τις συμφωνίες και χάνεται κάθε εναλλακτική άποψη. Συνειδητοποιείται λοιπόν ότι απομακρύνεται ε, πολίτες από τους ε, ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς με τρόπο που δεν κατάφεραν ο Φαράτς και η Λεπέν. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ξεκάθαρους όρους, έτσι είπατε, και αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα προς τους ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα της Επιτροπής μας, ή θα υποστηρίξουμε αγρότες ή ε, τις ε, συμφωνίες εμπορίου, όχι όμως και τα δύο. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευση. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος πολύ σημαντικής χώρας. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι, ευχαριστώ. Η μελέτη έχει πολύ αισιόδοξη προσέγγιση και προβλέπει θετικό αντίκτυπο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά οι παραχωρήσεις θα πρέπει να γίνονται με ανάλογο τρόπο, με συμμετρικό τρόπο ε, και οι προσβάσεις να είναι συμμετρικές ε, στις αγορές των τρίτων χωρών ενώ ε, φαίνεται ότι πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληρώνει με παραχωρήσει γεωργικών προϊόντων για να λάβει παραχωρήσει σε άλλου κλάδου. Και αυτό δυστυχώ δεν το λαμβάνει υπόψη η μελέτη. Επίση, η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει υποχρεώσει με βάση οικολογικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια ευημερία των ζώων και έχει και κάποιε υποχρεώσει λόγω τη προσπάθεια μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά, όλε αυτές οι πλέον υποχρεώσει αυξάνουν το κόστο παραγωγή. Λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη στις συμφωνίε με τις τρίτες χώρε καθόλου. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόιμπους. Okay, pani... Όχι, κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το παγκόσμιο εμπόριο ε, επηρεάζει και με ποιο τρόπο το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Γιατί Είμαι γιατρός και το, τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση των ε, ασθενειών του πολιτισμού, κυρίως αύξηση του καρκίνου. Ο καρκίνος και άλλες ε, αρρώστιες του πολιτισμού έχουν σχέση με την ε, μικροβιακή αντοχή και είναι αποτέλεσμα ακριβώς της δηλητηρίασης που έχουμε υποστεί από διάφορα προϊόντα. Εμείς έχουμε στην Πολωνία 300, 330 πρόσθετα στα τρόφιμα, χιλιάδες φυτοφάρμακα. Έχουμε τις ορμόνες, τις αυξητικές και άλλες ορμόνες που σε συνδυασμό με τα αντιβιωτικά αποδυναμώνουν το ανασωπητικό μας σύστημα. Και μάλιστα θα σταματήσουμε εμείς να παράγουμε αυξητικές ορμόνες, είπε κάποιος, όταν υπογράψουμε τη ΣΕΤΑ. Αυτό είναι αφελές αν μη τι άλλο. Δυστυχώς ε, το μόνο που ενδιαφέρει το εμπόριο είναι τα χρήματα. Κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ. Η μελέτη επικεντρώνεται στις εξαγωγές κυρίως ε, και στην προσπάθεια διεξόδων ε, εξαγωγικών από τις εμπορικές συμφωνίες και είναι θετικά τα αποτελέσματα για το γάλα όπως μας είπατε. Τι γίνεται όμως με την εσωτερική αγορά, γιατί ζητούμε θεμητό ανταγωνισμό ε, στη Γεωργία. Αλλά δυστυχώς ενέμεν ε, ναι, έχουμε πολύ πιο ποιοτικές παραγωγές, ε, αλλά έχουμε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες παραγωγής. Ενώ οι τρίτες χώρες ούτε αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές έχουν, ούτε κοινωνικές, ούτε υψηλά εργασιακά δικαιώματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ασφαλιστικές δικλείδες αποτελεσματικές για τα ευαίσθητα προϊόντα. Γιατί αλλιώ το κόστο θα πλήξει κυρίω και την ήθα την πληρώσουν οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Ερωτώ λοιπόν, πώ θα εξασφαλίσουμε την προστασία των γεωργών μα και να τους προστατεύσουμε από τον αθέμητο ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Επίσης, η εκτίμηση των ποσοστώσεων των εμπορικών συμφωνιών είναι σημαντική, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. άρα παραβαίνεται τη συνθήκη. Η κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια ερωτήματα. Για κάποιο λόγο η έρευνα της έσοδο στην Αμερική δεν χρησιμοποιήθηκε ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν τόσο πολλοί τομεί, όπως είναι το, για παράδειγμα ε, το ε, μέλι. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε το επίπεδο που μπορεί να φτάσει η ανάπτυξη. Επίσης λοιπόν, ε, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα καθυστέρησης, αναλύσεις, τι συμβαίνει με το χοιρινό κρέας ε, και ούτω καθεξής για ποιο λόγο οι αποδόσεις ε, των αγροτών δεν έχουν συμπεριληφθεί οι επιθυμίες ε, της κοινωνίας προς την ε, γεωργία δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτή η έρευνα έχει ε, ελλείψεις, δεν έχει οικονομικές αναλύσεις, το ζήτημα δεν αφορά την κοινωνία, αφορά μονάχα το εμπόριο και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος διότι δεν αφορά την κοινωνία, για σας σας απασχολεί μονάχα το εμπόριο και επίσης ποιος συνέταξε αυτή την έρευνα θεωρεί ότι η σχέση εμπορίου και αγροτικών προϊόντων είναι το ίδιο με τη γεωργία. Η γεωργία όμως και το εμπόριο τέτοιων προϊόντων είναι δύο διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό το λόγο θα χάσει η γεωργία μας διότι εσείς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε αυτή τη διαφορά. Ο κύριος Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω πόσο σημαντικές μπορεί να θεσυφωνεί στην οικονομική ανάπτυξη έχουν με κάποιες χώρες όπως Εκουαδόρ και άλλες, αλλά εκπροσωπώ την Νότια Ιταλία εδώ και ανησυχώ από τη μελέτη όσον αφορά τις ορευτικά αποτελέσματα 12 μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών για τον αγροτροφημικό τομέα. Συνοπτικά θα καταλάβω ότι πρέπει να εξηγήσουμε στους γεωργούς μας που αυτά τα χρόνια εκμεταλλεύτηκαν ε, με τις αρνητικές συνέπειες των συμφωνιών με τις χώρες της Βορείου και δεν μπορεί να ανταγωνιστική σε μια αγορά που κυριαρχείται στι πολυεθνικές. Και μειώνουν μέσω των συμφωνιών οι πολυεθνικές την τιμή της παραγωγής. Τι να πούμε στους γεωργούς που τους καθησύχασα οι διάφοροι πολιτικοί στην Ιταλία ε, για τη ρήτρα διαφύλαξη των ενεργοποίηση που προβλέπεται στις συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες Βορειοαφρικής κάτι που δεν έγινε ποτέ απαντούμε μελέτη αντικτύπου που δεν έχει ενδελεχή μελέτη για όλα τα γεωρικά προϊόντα. Και από την εξολόγηση εξαιρεί τους ευάλωτους τομείς. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Αυτό θα ήθελα ξεκάθαρα να γνωρίζω από αυτές τις συμφωνίες. Εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Ε, ξέρω κύριε Επίτροπε ότι βιάζεστε και λυπούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα δώσω πρώτα σε εσά το λόγο, κυρία Μάλμστρομ. Σας ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι η μελέτη που σας παρουσιάσαμε έχει και κάποια όρια. Και ήμουν ειλικρινής από την αρχή γι' αυτό. Ε, ίσως λόγω έλλειψη μεθοδολογίας, λόγω πείρας, γιατί υπάρχουν πάντα κάποια πρίσματα που χρησιμοποιούμε, αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε τέτοιε μελέτε όταν συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίε και κυρίω δίνουμε έμφαση σε κάποιου ευαίσθητου τομεί. Και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτέ τι ευαισθησίε. Και είναι μία από μία σειρά μελετών, αλλά αναγνωρίζω ότι έχει τα όρια τη και ίσω τις πιο λεπτομεριακέ ερωτήσει, θα τι απαντήσει ο επίτροπο Χόγκαν. Οι εμπορικέ συμφωνίε χρειάζονται για την οικονομική μα ανάκαμψη. Γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε με τις αγορές που έχουν υψηλή ανάπτυξη εκτός της Ευρώπης και οι εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν δεν είναι πανάκια, δεν λύνουν όλα τα οικονομικά προβλήματα, δεν δίνουν απαντήσεις για τα πάντα, αλλά έχουμε βάσιμες αποδείξεις ότι ε, δημιουργούν πρόσφορα έδαφος για δημιουργία θέσης απασχόλησης και για επενδύσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι για όλους και όχι με ισότιμο τρόπο για όλους και σίγουρα δεν είναι πανάκι από μόνε του για την οικονομική μα κρίση. Θα πρέπει να συμπληρωθούν με άλλε οικονομικέ δραστηριότητε. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε τέτοιου είδου εκτιμήσει και απολογισμού. Για να δούμε πού έχουμε ευάλωτου τομεί, ώστε από την αρχή να μετριάζουμε τα αρνητικά αποτελέσματα σε αυτού. Και ε, αυτές οι προσβολές ε, και, οι, και μοφές για νεοφιλελευθερισμό και τραμπισμό δεν ευνοούν το διάλογο. Εγώ ήρθα εδώ για διάλογο. Θέλουμε μια εμπορική πολιτική, περιεκτική, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή, που αναδράζεται σε αξίες. Μπορεί να μην συμφωνείτε και συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποιοι χαμένοι από την παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να κάνουμε πολύ περισσότερα ώστε να μετριάσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο τις, τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης για να είναι έτοιμος ο κόσμος αλλά δεν πρέπει να κατηγορείτε τις εμπορικές συμφωνίες ε, για όλα τα κακά του κόσμου και για την απόλυτη θέση απασχόληση. Που μερικέ φορέ η απόλυτη θέση απασχόληση οφείλεται στην τεχνολογική ανάπτυξη. Βέβαια, αυτό δεν ενδιαφέρει ε, του ε, πολίτε. Ε, ο, κύριος πολι... Οι πολίτε ενδιαφέρονται για σωστέ ε, συμφωνίε. Και κύριε Δαραμπέλα, δεν έχουμε συμφωνία με τη Σενεγάλη, κακώ μα κατηγορείτε. Έχουμε συμφωνίε ε, με κάποιε περιφέρειες τη ε, Αφρική, ασυμμετρικέ. Ανοίγουμε περισσότερε αγορέ μα και θέλουμε άνοιγμα του. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάποιου ευάλωτου τομεί. Έχουμε στενή συνεργασία με το επιτελείο του Επιτρόπου Μίμητσα για την ανάπτυξη, γιατί θέλουμε να συμβαδίζουν το εμπόριο με την ανάπτυξη. Και έχουμε και στρατηγική περιφερειακή ολοκλήρωση. και μάλιστα οι Αφρικανικέ χώρε που συνήψαν συμφωνίε σε εταιρική σχέση μαζί μα ε, ε, ήταν ενθουσιώδει για αυτές και έχουμε στενή συνεργασία με τι κυβερνήσει τι Αφρικανικέ, ε, που πέτυχαν και την έγκριση των κοινοβουλίων του, κάτι που είναι πολύ θετικό. Με τη Σενεγάλη δεν έχουμε αντίστοιχη συμφωνία. Μου αναφέρατε παράδειγμα τον Τακάρ, θα το ελέγξω. Αλλά αυτή τη φορά τουλάχιστον δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασία ή άμυνα στο εμπορίο, προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε και να τα ε, επικαιροποιήσουμε για να αντιμετωπίζουν ε, αποτελεσματικά τις απειλέ και καλύπτουμε και το dumping στη Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τα, τα εξαγωγικά στοιχεία, τα έχουμε, όχι εδώ, όχι μαζί μου, αλλά ε, μπορούμε να σα στείλουμε λεπτομεριακά στοιχεία για τι εξαγωγέ τη κάθε χώρα. Κυρία Ρενά, για τις ε, μεγάλες εταιρείες που είναι κερδισμένες. Ναι, όντως είναι πολλές μεγάλες εταιρείες που βρέθηκαν κερδισμένες, αλλά και μικρομεσαίες επίσης επωφελήθηκαν. Και έχω και παραδείγματα. Και για τις συμφωνίες με το Περού και την Κολομβία, από τότε που τέθηκαν σε ισχύ, 1.500 ε, ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις άρχισαν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Περού και το ίδιο και από την πλευρά του Περού. Εκατοντάδες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, επίσης της Κολομβίας άρχισαν να δραστηριοποιούνται χάρη στις συμφωνίες αυτές και έχω τα στοιχεία που είναι πρόσφατα και είναι και πολύ θετικά τα νέα αυτά. Αυτά κύριε, κύριε Πρόεδρε, βάζω τελεία εδώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και αν κάποια στιγμή ε, αισθανθήκατε ότι σας προσβάλαμε, σας ζητώ Συγγνώμη, Σίγουρα δεν ήταν η πρόθεσή μας να σας προσβάλλουμε. Και τώρα, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πρέπει σε λίγο να τελειώσουμε. We don't conclude agreements at any cost, Mr. Zulu. Πιστεύω ότι αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική διότι μας ε, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα διάφορα ε, σενάρια τα οποία έχουμε εξετάσει σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικές πληροφορίες που ε, λαμβάνουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή. Στην μελέτη σίγουρα οι περισσότεροι διάβασαν την περίληψη αν ε, το κάνατε αυτό ε, θα βλέπατε ότι οι παράμετροι ήταν ε, πιο αναλυτικοί. Κάναμε δύο τεχνικά μοντέλα για μία έρευνα και δεν συμπεριλαμβάναμε κάποιες υποθέσεις διότι δεν, δεν συμφωνούμε με τις υποθέσεις. Δεν θεωρούμε ότι είναι έγκυρες όμως ε, για να μπορέσω να βοηθήσω όσους ενδιαφέρονται πραγματικά θα, θα αποστείλω μία επιστολή σε όλα τα μέλη των δύο επιτροπών όπου ε, θα δίνουμε περισσότερες προφορίες μέσα σε μία ε, σελίδα για όσους δεν έχουν διαβάσει όλη τη σελίδα, όλο το κείμενο διότι 32 χρόνια πολιτικός ξέρω πώς γίνεται η όλη δουλειά. αναφερθήκατε ε, σχετικά με το όφελος ε, των αγροτών και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε εμείς ως Επιτροπή να ε, αντιμετωπίσουμε και έχουμε το διεθνές εμπόριο το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν θα βασιστούμε με, στα αποτελέσματα του Task Force και θα σας ενημερώσουμε το 2017 για το συγκεκριμένο θέμα για να δούμε τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε καθώς επίσης ε, και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο τόνισα ήδη από τις ακροάσεις μου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τη βοήθεια άλλων γενικών διευθύνσεων ανταγωνισμού, λό, νόμου, δικαίου ε, και να κάνουμε κάποιες προτάσεις το 2017. Και συμφωνώ επίσης με, τον, ε, κύριο με την κυρία Γκρεσέ ότι χρειαζόμαστε αμοιβαιότητα. Χρειάζονται δύο για να χορεύσουν γκο η φλαμίγκο στη δική σας περίπτωση. Και συμφωνώ απόλυτα με εσάς και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό όσον αφορά ε, ζητήματα ε, των ε, φυτών, ε, κυρία Μαρίνο, έχουμε κάποιες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με τους εταίρους μας στη Βόρεια Αφρική και υπάρχουν έλεγχοι στα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτά τα ζυζανιοκτώνα να φτάσουν και αυτές τις ασθένειες να φτάσουν στην Ευρώπη. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να έχουν να προσέχουν και να εφαρμόζουν τους σωστούς ελέγχους διότι ε, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για οτιδήποτε πηγαίνει στραβά. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι υπεύθυνα πάνω σε αυτό και εμείς ε, θα συνεισφέρουμε σε αυτό για να γίνει σωστή δουλειά. Και ε, όσον αφορά την κυρία Κούπερ, εργαζόμαστε ε, στο ζήτημα το οποίο προεργαμβάνεται στην διακήρυξη G20 για την Γεωργία. Είναι μια πρόοδος, όμως έχουμε να διανύσουμε ακόμα μεγάλο, ε, μεγάλη απόσταση όσον αφορά τα ζητήματα των ζυζανιοκτώνων. Και εδώ φυσικά υπάρχει και το ζήτημα των εισαγωγών, ε, το οποίο θα είναι και το πόσο αυτό θα υποφελεί στο περιβάλλον. Ο κύριος Σταρτάν ανέφερε ε, το βοδινό κρέας, ναι, εάν ένα τέτοιο σενάριο, ε, συμφωνούσαμε πάνω σε αυτό, τι θα συνέβαινε αν αναλογιζόμασταν τι συνέπειες όλου αυτού. Ναι, είναι χρήσιμο για όλους εμάς ε, να το κατανοήσουμε, όπως είπε η κυρία Μάλμστρομ. Όμως η βάση περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και σε αυτό θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή και αυτά είναι μονάχα σενάρια. Δεν προτείνουμε, δεν λέμε ότι θα εφαρμοστούν, απλά σας λέμε ποιες θα είναι οι συνέπειες στα διάφορα σενάρια, τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που συμφωνούσαμε. Και κύριο κύριε, όσον αφορά την Ιδονησία οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ καλές και στην περιοχή ΑΖΕΑΝ υπάρχουν 750 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ε, στην Ινδονησία παίρνουν τα προϊόντα τους κυρίως από την Αυστραλία ε, και υπάρχει 25% ε, αυτονομία για κάποια προϊόντα, όμως υπάρχει δυνατότητα για ευρωπαϊκές εταιρείες ε, να δραστηριοποιηθούν στην Ινδονησία αλλά και στο Βιετνάμ και εκεί συζητούμε για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όμως θα χρειαστούν χρόνια για να ολοκληρωθούν, όμως παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Η εικόνα, κύριε Τσέλεμπερα δεν θα είναι καλές αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτά τα σενάρια. Η κυρία Μάνστρον απάντησε ε, στις ανησυχίες σας, ε, κύριε Μαγκίνη, σχετικά με το τι θα κάνουμε. Η συνέπεια της έρευνας είναι ότι απλά ενημερώνει και ήδη υπάρχουν ε, τα μέσα ελέγχου Κυρία Αγγιλέρα, συμφωνώ πολύ με εσά ότι οι αγρότες έχουν δυσκολίες, όμως θα πρέπει να διαχειριστούμε την αγορά με βάση την ε, προσφορά και τη ζήτηση και αφού γίνει αυτό, στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν επαρκεί για τους αγρότες, όμως κατευθύνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν μεσογειακά προϊόντα όπου θα πρέπει να κάνουμε ένα περαιτέρω έλεγχο για να δούμε τις συνέπειες και ε, όσον αφορά προϊόντα όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, εκεί θα σας δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Κύριε Ντότς, ε, αυτό που είπατε και ε, το Brexit, δεν πρόκειται τώρα το απόγευμα να διαπραγματευτούμε το Brexit. Δεν θα το κάνω ούτω ή άλλω και αργότερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε μία απόφαση να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διώξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εσεί μόνοι σα το αποφασίσατε. Και ίσω δεν έχετε σκεφτεί όλε τι συνέπειε πολύ σωστά. Ελπίζω να τι εξετάσατε όλε τι συνέπειε πριν λάβετε αυτή την απόφαση. Μακάρι. Πάντω, ε, γνωρίζω ότι έμειναν ε, εκρεμεί πολλά ερωτηματικά και η κυρία Φλάναγκα, σίγουρα υπάρχουν ε, διαφορέ αγιαφύρωτε μεταξύ μα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι θετική η συμφωνία για, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρω πώ ασχολείστε με τα περιβαλλοντικά και για την προστασία και θα εξετάσετε πολύ θετικά τα θετικά βήματα που έγιναν για το περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ε, ευημερία των ζώων, ε, εργασιακές προδιαγραφές που αναφέρονται πολύ ε, ρητά στη συμφωνία είναι οι υψηλέ προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι οποίε είμαστε υπερήφανοι και πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Αυτά πρέπει να ολοκληρώσω. Θα σα υποβάλω και σημείωμα και στι δύο ε, με τη σύνοψη, πιο εκτεταμένη σύνοψη τη μελέτη που εκπονήσαμε. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε, περιμένουμε και γραπτό τι ε, πληροφορίε αυτέ. Ήταν πολύ θετική αυτή η ανταλλαγή απόψεων ε, και μην ξεχνάτε ότι οι βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας έχουν άμεσες επαφές με τους γεωργούς και σας μεταφέρουν εδώ τις αντιδράσεις τους ε, και την αίσθηση που έχουν από την όλη συζήτηση. Και σας παρακαλώ μην ξεχνάτε τη γεωργία στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Και τελευταίο θα λάβει το λόγο ο συμπρόεδρος, ο πρόεδρος της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ε, Βεβαίω, έχουμε πολύ καλή συνεργασία οι δύο επιτροπέ Γεωργία και Διεθνού Εμπορίου. Πολύ καρποφόρα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και καλό σας βράδυ. Ε, σας ευχαριστούμε και εμείς και επιβεβαιώνουμε και εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Εμείς θα ξανασυνδυθούμε στις στις 5 Δεκεμβρίου και ευχαριστώ για τους διερμηνείς για την ε, υπέρβαση του εμπορίου και εύχομαι, ε, και εύχομαι καλό σας βράδυ.